Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich Συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είναι δύσκολη η Δευτέρα το απόγευμα γιατί όλοι ταξιδεύουν, αλλά είμαστε ακόμα πολύ άρεθμοι, πολύ περισσότεροι από την προηγούμενη Δευτέρα τέτοια ώρα. Και αυτό φυσικά είναι αυτονόητο γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Να ακολουθήσουμε όμως την ημερήσια διάταξη. Έχετε μπροστά σας την έγκριση. Για τους συντονιστές να πω ότι δεν θα συνεδριάσουμε σήμερα στις 6, αλλά αύριο στις 8.30. 8.30 ακριβώς για να ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη αύριο στις 9. Έχουμε μπροστά μας και τις κάμερες που τραβάνε και έχουμε και τους επισκέπτες μας, τη συναδέλφου Λίχτενμπεργκ από την Αυστρία. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή Προϋβάλλοντος. Δεν έχουμε ανακοινώσει του Προέδρου. Και γρήγορα γρήγορα να περάσουμε στο σημείο 4, λέει ο Πρόεδρος, μάλλον το σημείο 3. Ανταλλαγή απόψεων με την Κόνη Χέντεγάρτ, την Επίτροπο για την Κλιματική Αλλαγή. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Χέντεγκάρντ. Φυσικά είναι κορυφαία σημασία στο θέμα της αλλαγής του κλίματος και μας ε, απασχολεί όλους, γι' αυτό είναι και τόσο αθρώα η προσέλευση. Σήμερα έχουμε την τελευταία μεγάλο γύρο των κρατών μελών στην Κίνα για την προετοιμασία του κόπου το Κανκούν. Δεν γνωρίζουμε ασφαλώς τι θα προκύψει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας για τη θέση μας για το Κανκούν, για τη δική μας τοποθέτηση και το Νοέμβριο θα περάσει στην Ολομέλεια το θέμα αυτό. Θα ασχοληθούμε επίσης με τις ανακοινώσεις σας για το 20% μέχρι το 2020 σε ό,τι αφορά τις εκπομπές του άνθρακα, συν. Αυτό το 20% συν θα το διευκρινίσουμε. Διάβασα την, ε, την γερμανική εφημερίδα και βρήκα αυτή την όμορφη φωτογραφία της κυρίας Χέντεκαρτ με την εξής επιγραφή ότι η Επιτροπός Κόνη Χέντεγκαρτ θέλει μέχρι το 2020 να μειώσει περαιτέρω α, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα πέρα από το συμφωνηθέν 20%. Άρα σας δίνω το λόγο πάρα αυτά για να συζητήσουμε τις εξέλιξεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα για την ε, συνάντηση αυτή και σκοπός αυτού του διαλόγου είναι να καταφέρουμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες και από εσά τους ευρωβουλευτές. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι θα είμαι πολύ σύντομη στην αρχική μου παρέμβαση. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε και εσείς στη συνέχεια να πάρετε το λόγο, να θέσετε ερωτήσεις. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, να μιλήσω για ένα μισάωρο δηλαδή, προτιμώ να είμαι σύντομη στην αρχική μου παρέμβαση. Όπω ξέρετε, στην παρουσίαση για την κατάσταση Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και το σημείο αυτό ήταν το σημαντικότερο, θέλετε, ζήτημα στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες επενδύσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση και οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα παραμείνει μαζί μας για τα επόμενα χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μία μακρόπνοη πολιτική. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ έντονη, είδαμε στο παρελθόν, ε, με συγχωρείτε, μια πολύ στο παρελθον οικονομική ανάπτυξη, η οποία όμως οδήγησε σε μια μη βιώσιμη κατανάλωση των ε, πρώτων υλών, καθώς επίσης και των ορυκτών καυσίμων. Το ζήτημα αυτό απασχόλησε πολύ τις κυβερνήσεις και είδαμε ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, προκειμένου να έχουμε μια υφόρο, βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ε, στην επιστολή προς τον πρόεδρο Μπούζεκ, ο πρόεδρος Μπαρόσο τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πιο συντονισμένη δράση της στρατηγικής μας για το 2050, επίσης το ενεργειακού χάρτη για το 2050 και τη στρατηγική που ακολουθούμε για τις μεταφορές. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συγκεράσουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες με έναν τρόπο συνεκτικό, προκειμένου να μην δρούνε τελικά κατακαιρματισμένα, αλλά με έναν τρόπο πολύ πιο ευθυγραμμισμένο και συντονισμένο. Να, είναι λοιπόν η σημαντική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε το πακέτο μέτρων για την κλιματική αλλαγή και για την ενέργεια και γι' αυτό η εφαρμογή του πακέτου αυτού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του προγράμματος για το 2011 λαμβάνονται κάποια συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής, όπως για παράδειγμα το μέτρο ε, εμπορίας των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, που χρησιμοποιείται ε, ένα σύστημα πληστηριασμού. Καθώς επίσης και το ότι θα πρέπει το σύστημα αυτό, το ETS, να εφαρμοστεί, σύστημα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και αποτελεί σημαντική πρόκληση για αυτά. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε τρεις στρατηγικές πρωτοβουλίες για το 2011. Πρώτον, τον έχουμε έναν ενεργειακό χάρτη με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα με 2030, Επίσης, να καταφέρουμε να περάσουμε ενεργειακές πολιτικές, και για την κλιματική αλλαγή σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπειτα η συνέχιση των διαπραγματεύσεων μετά το Κανκούν. Τα πρώτα δύο στοιχεία εντοπίστηκαν στην παρέμβαση του κυρίου ε, Μπαρόσο και το τρίτο θα το δούμε περισσότερο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το Κανκούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να δίνει μία μάχη σε εσωτερικέ και εξωτερικές πολιτικές της για τις κλιματικές αλλαγέ. Θέλουμε να προωθήσουμε ένα, από τα πιο φιλόδοξα παγκοσμίως προγράμματα για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και να καταλέξουμε επίσης σε μια παγκόσμια συμφωνία προκειμένου να μειωθούν παγκοσμίω οι εκπομπές διοξείδου του άνθρακα. Όσον αφορά τον οδικό χάρτη 2050 για μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξίου του άνθρακα. Το πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τις επόμενες αλλαγές είναι σημαντικό να καταφέρουμε να περάσουμε πέρα από το στόχο μας της μείωσης του 20% και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε ένα μακρόπνο δικό χάρτη για μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και επίσης να αρχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε και τους στόχους για το 2030. Οι στόχοι του 2030 θα αποτελέσουν κατευθυντήρια γραμμή για τη συζήτηση που γίνεται για την στρατηγική Ευρώπη 2020. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους του 2030, δεν μπορούμε να μην δραστηριοποιηθούμε μέχρι το 2020. Όλα αυτά θα αποτελέσουν λοιπόν τμήμα του προγράμματος εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 και θα ακολουθήσουμε όλα τα ενδιάμεσα βήματα μέχρι να φτάσουμε τους στόχους του 2020 και του 2030. Στην ανακοίνωση που έγινε τον Μάιο, δόθηκε η βάση προκειμένου να γίνει μια περαιτέρω συζήτηση για τα ζητήματα αυτά. Τα ζητήματα συζητήθηκαν πλήρως στο Συμβούλιο και αντικατοπτρίζονται σε μία έκθεση του Προέδρου που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος την επόμενη εβδομάδα. Προσβλέπουμε επίσης την αντίδραση και τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να δούμε πώς, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλλει περισσότερο με το πρόγραμμα εργασίας του 2011 προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να πετύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους της. Οι κλιματικές αλλαγές ε, επηρεάζουν ε, πάρα πολλές πτυχές της οικονομίας και της κοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υπηρεσίες υγείας, την γεωργία, τις μεταφορές, την αλία, τα οικοσυστήματα, καθώς επίσης και τις υποδομές. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί οι οποίοι επηρεάζονται από αυτά τα οποία κάνουμε εμείς στον τομέα της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι τομεί να γίνουν πιο ανθεκτικοί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και να καταφέρουν να συμβάλλουν στην γενικότερα πιο ανθεκτική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να ταποκριθούμε στι προκλήσει αυτέ, θα πρέπει οι πολιτικέ για, την Ευρω... για την κλιματική αλλαγή να περάσουν, να αποτελέσουν τμήμα όλων των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουμε δηλαδή μια οριζόντια προσέγγιση. Είναι σημαντικό να γίνονται οι απαραίτητε εκθέσει προκειμένου να μπορούμε να αξιολογούμε αν όντω οι στρατηγικές μας και οι πολιτικές μας από το 2013 και μετά ευθυγραμμίζονται στο στόχο των κλιματικών αλλαγών. Επίσης έχουμε και την γενικότερη στρατηγική Ευρωπαϊκή 2020, η οποία και αυτή με τη σειρά της αναφέρεται στο ότι θα πρέπει να γίνει πιο ανθεκτική η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κλιματικές αλλαγές και ότι θα πρέπει να τεθούν οι απαραίτητοι στόχοι προκειμένου να προσαρμοστούμε περισσότερο στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών. Να αφαιρθώ επίση και στον προπολογισμό αυτή τη στιγμή, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον εξυγχρονισμό του προπολογισμού μα προκειμένου να θέσουμε τι απαραίτητε προτεραιότητε για την ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 συμπεριλαμβανομένη της πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγές. Το επόμενο πλαίσιο δημοσιονομικών πολιτικών θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης θέλουμε να θέσουμε ως προτεραιότητα μια ξεχωριστή νομική βάση για χρηματοδότηση προγραμμάτων κατά των κλιματικών αλλαγών. Δυστυχώ η Επιτροπή Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψε την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ουσιαστικά ήθελε να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στον υφιστάμενο προπολογισμό και το νέο μέσο χρηματοδότηση το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε και ελπίζω ότι θα διορθωθεί η στάση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα καταφέρουμε να βρούμε την κατάλληλη λύση. Επίση, θέλουμε την κατάλληλη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να πετύχουμε και τη χρηματοδότηση μελλοντικών πρωτοβουλειών στου μελλοντικού προπολογισμού. Νομίζω ότι θα κερδίσουμε θα καταφέρουμε να αποφεληθούμε πολύ αν δημιουργήσουμε τους απαραίτητους στόχους και δημιουργήσουμε ξεχωριστές γραμμές για την κλιματική αλλαγή στον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ο τομέας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συντονισμό στο τι κάνουμε στο μέλλον. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μιλήσω πολύ για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όπως είπε και ο πρόεδρος πριν από λίγο, γίνονται αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις στην ε, Κανκούν, Γίνονται διαπραγματεύσει με συγχωρείτε στην Κίνα, οι οποίε προηγούν και πραγματεύσεων που θα γίνουν στο Κανκούν. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα συνεδριάσαμε στη Νέα Υόρκη. Πριν από μερικέ μέρε έγινε μια υπουργική διάσκεψη στη Νέα Υόρκη με την ε, παρουσία πολλών υπουργών περιβάλλοντος και υπουργών ε, για την κλιματική αλλαγή και το βασικό μήνυμα της διπουργικής αυτής συνδιάσκεψης ήταν ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις που γίνονται στην Κίνα να καταφέρουν οι αρμόδιοι από το κείμενο αυτό των 75 σελίδων που έχουν μπροστά τους να εντοπίσουν τους τομείς εκείνους όπου χρειάζονται μεγαλύτερη πολιτική καθοδήγηση προκειμένου να καταφέρουν να καταλήξουν σε μια φιλόδοξη συμφωνία. Μεταξύ λοιπόν του Τσίντσιν και του Κανκούν οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί θα πρέπει να ταποκριθούν σε αυτές τις πολιτικές προκλήσεις και θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα εκρεμή ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί ακόμα. Ξέρετε ακόμα και φάνηκε αυτό και στην Κοπενχάγη ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή μπορούν να επιτευχθούν πολύ σημαντικά πράγματα. Επομένω είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε σε πραγματεύσει αυτέ που γίνονται προπαρασκευαστικά αυτή τη στιγμή μέχρι να φτάσουμε στο Κανκούν. Θα επανέλθουμε προφανώς στο σημείο αυτό. Ένα άλλο τομέα που πρέπει να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη είναι πώ μπορούμε να καταφέρουμε να μιλήσουμε όλοι με μία ενιαία φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα αυτό είναι και παραμένει πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που βλέπουμε ότι δεν μιλά η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία ενιαία φωνή. Το χρειαζόμαστε πάντως αυτό, είναι απαραίτητο και θα πρέπει και εσεί, ω ευρωβουλευτέ, να αποστείλετε πιο ξεκάθαρα το μήνυμα αυτό προ τα έξω και ιδίω εν του Κανκούν. Εν κατακλείδη να αφαιρθώ πολύ σύντομα σε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες ένας τομέας είναι ενδεχομένως η χρησιμοποίηση μιας νέας έκθεσης και καταγραφής της χρήσης της γης, πώς μπορεί το σύστημα αυτό να ενσωματωθεί περισσότερο στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Δεν καλύπτεται ακόμα η χρήση της γης στο Ευρωπαϊκό ETS. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν πει ότι όλοι οι τομείς θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο ETS και υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι ακόμα δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Επίσης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναρμονισμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μολονότι οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Κλιματική Αλλαγή προβλέπουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ευθυγράμμιση. Χρειάζεται ανάληψη δράσεων σε πάρα πολλούς τομείς προκειμένου όντως ε, το σύστημα αυτό να εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρξει ε, μια ε, ισότιμη παρακολούθηση και καταλογισμός χρηματοδότησης από όλα τα κράτη-μέλη. Το 2011 λοιπόν θέλουμε να υποβάλουμε μια έκθεση που θα περιλαμβάνει και μια αξιολόγηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης του προγράμματος της, των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, για το 2020 προβλέπονται νέες διατάξεις όσον αφορά την υποβολή αναφορών, υποβολή εκθέσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της στρατηγικής του 2020 και λέμε επίση ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση, για παράδειγμα. Και επίση θα πρέπει να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε στη δική μας νομοθεσία τις απαιτήσει προβλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη για υποβολή εκθέσεων και αναφορών για την κατάσταση του περιβάλλοντο. Επαιτείται λοιπόν από τα κράτη-μέλη μεγαλύτερη συμμετοχή μεγαλύτερη ενσωμάτιση τη κοινοτική νομοθεσία στην εθνική νομοθεσία, καλύτερη επιβολή τη νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξάλληψη οποιοδήποτε, γραφειοκρατικού άκθου που θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην εφαρμογή τη κοινοτική νομοθεσία για τι κλιματικέ αλλαγέ. Επίσης, γίνεται ήδη μια αξιολόγηση της εφαρμογής της ε, Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την αξιολόγηση που θα γίνει αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια νέα έκθεση που θα βασίζεται σε αυτή την αξιολόγηση. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα πράγματα για το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε όμως ότι πάρα πολλές από τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε για τις κλιματικές αλλαγές του 2011 περνάνε μέσα από διάφορους τομείς όπως η ενέργεια, όπως οι μεταφορές. Και το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να συνεργαστούμε είναι πώς θα καταφέρουμε να προσαρμόσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές, που θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση για την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση των ιδέων αυτών. Όντως η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία του κλίματος θα πρέπει να ενταχθεί και στις άλλες πολιτικές. Μόνο έτσι θα πετύχουμε και έχουμε πριν από κάποιες εβδομάδες λάβαμε μια πρόταση για την μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής και εκεί θα ξεκινήσουν τα πράγματα γιατί είναι πολύ σημαντικό ο τομέα αυτός για την ε, άλλαγη του κλίματος. Μετά θα έχουμε τα διαρθρωτικά ταμεία, αναφέρατε την ε, μέσοπρόθεσμη διαμόρφωση της χρηματοδότησης θα πρέπει να συμμετάσχει και σε αυτή την πολιτική η αλλαγή του κλίματος για να μην περιοριστεί σε έναν μόνο τομέα. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο, πάνω από 20 άτομα, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σας περιορίσω τρία λεπτά για τους συντονιστές και θα δούμε τι θα γίνει για τους υπόλοιπους. Ο κύριος Ζήμπρα το λέω Καταρχάς ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο για την ε, σημαντική της δέσμευση και νομίζω ότι το mainstreaming ασφαλώς αποτελεί το βασικό στοιχείο για να πετύχουμε στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος. Ξέρω ότι είναι πολύ ρεαλίστρια η Επίτροπο σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες από το Κανκούν σε σχέση με την Κοπενχάγη. Θέλουμε να υπάρξει νομικά δεσμευτική ε, συμφωνία. Αν δεν την πετύχουμε αυτή, δεν θα είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Αλλά κυρία Επίτροπε, ποια θεωρείτε ότι είναι τα συγκεκριμένα ορόσημα για να κρίνουμε κατά πόσον θα έχει αποτύχει ή θα έχει πετύχει το Κανκούν. Συγκεκριμένα, πείτε μας τι προσδοκάτε, τι θεωρείτε ότι θα καθορίσει κατά πόσο πέτυχε ή μη το Κανκούν σε σχέση με την προσέγγιση των ΗΠΑ και της Ευρώπης. κοιτώντα θέματα mainstreaming νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία εδώ στα αντιρρετικά ταμεία σε ό,τι αφορά τη θερμομόνωση προκειμένου να βελτιωθεί η εξοικονόμηση ενέργειας. Ποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναλυφθούν και όπως ξέρουμε δεν ε, είναι πολύ ικανοποιητική η κατάσταση με τα κτίρια σε ό,τι αφορά τη θερμομόνωση σε όλη την Ευρώπη. Και εδώ λοιπόν θα χρειαστούν πρωτοβουλίε. Άλλη μία ερώτηση για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ξέρετε ότι ως Επιτροπή λάβατε την ε, εντολή να κάνετε προτάσεις για νομοθεσία για τα προϊόντα. Για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια σε ό,τι αφορά το φωτισμό. Και αυτό σε πολλές χώρες έχει προκαλέψει ε, μεγάλες αντιδράσεις σε ό,τι αφορά τους λαμπτήρες, για παράδειγμα. Πότε όμως ε, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπε προτάσεις για τη μεγαλύτερη οικονομική, ενεργειακή συγγνώμη, αποδοτικότητα. Γιατί με το φωτισμό έχουμε καλύψει μόνο ένα τομέα. Ευχαριστώ, Κυρία Ζέιμπερ, ο κύριος Γιώργενσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την ε, Επίτροπο Χίριγκαρτ. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες ε, προφανώς συμφωνούμε όταν λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει την ηγεσία της. Ωστόσο, κοιτώντας την κατάσταση και πώς έχει αλλάξει μετά την Κοπενχάγη, πρέπει να πούμε ότι η κατάσταση δεν έχει ουσιαστικά μεταβληθεί. Μας ε, κάνατε μια ανακοίνωση και είπατε ότι πολλά μπορεί να γίνουν για να υπάρξει μείωση των εκπομπών. Και ναι, όντως πραγματικά, αν γίνουν όλα αυτά, έχουμε ευκαιρία να αναλάβουμε την ηγεσία. Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε επίσημη απόφαση. Εξακολουθούν να ακούγονται φωνές ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τον στόχο του 20% και να μην πάμε παραπέρα. Άρα, σας ρωτώ, πότε θα έχουν διαμορφωθεί η σωστοί όροι και εμεί θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει όχι μόνο γιατί θα περιοριστεί η αλλαγή του κλίματος, αλλά γιατί θα τονωθεί και η ανταγωνιστικότητά μας. Και τελευταία ερώτηση. Πώς μπορούμε να διτηρήσουμε την αξιοπιστία μας έναντι των πιο φτωχών χωρών του κόσμου, αν εμείς οι ίδιοι δεν τηρούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για να πετύχουμε να μην αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από 2, βαθμούς. Είναι πραγματικά παράλογο το ότι γίνεται. Ευχαριστώ που μίλησατε αγγλικά, λέει ο πρόεδρος, ο Κρις Ντέιβις. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Νομίζω, επίτροπε, ότι δεν έχετε αναλάβει το αξίωμά σας σε μια καλή συγκυρία, γιατί δεν είναι πολύ δύσκολοι όροι. Κοιτώντας το Κανκούν, προφανώς λείπει η πολιτική βούληση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φυσικά έρχεται και η Κίνα και η Ινδία, αλλά έχω την εντύπωση ότι ακόμα περιμένουμε από τις ΗΠΑ να αναλάβουν την ηγεσία. Η είπα με την ε, πιο υψηλή, το πιο υψηλό ποσοστό εκπομπών κατά κεφαλή την πιο μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη. Χωρίς τη ΣΥΠΑ δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε διεθνή συμφωνία και φυσικά επί του παρόντο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι η ΣΥΠΑ πρόκειται να αναλάβουν τα ενία αυτά. Όλο και πιο δύσκολο καθίσταται να πετύχει το οτιδήποτε, να περάσει το οτιδήποτε ο πρόεδρος Ομπάμα από το Κογκρέσο. Αν θα θέλετε να σχολιάσετε παρακαλώ. Και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε δίκιο ότι θα πρέπει να ενταχθεί η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και στις υπόλοιπες πολιτικές. Νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό παράδειγμα. Έγινε μια συζήτηση πέρσι, την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη, για τη μείωση των εκπομπών σε ό,τι αφορά τα ελαφριά εμπορικά οχήματα. Φυσικά ε, γίνεται και πολύ lobbying κατά της πρότασης αυτής και αν θα παρουσιαστεί ως ε, project μέτρο κατά αποτελεσματικότητα των καυσίμων και όχι ως μέτρο μείωσης ε, του διοξιδίου του άνθρακα, θα ήταν εύλογη αυτή η αντίδραση. Αλλά προς το παρόν θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και τι θα ψηφίσει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα παρουσιάσουμε κάθε πολιτική για να δράξουμε τα μέγιστα ωφέλη, όπως είπατε. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τις αμφιβολίες, το σκεπτικισμό που επικρατούν για την αλλαγή του κλίματος, νομίζω ότι η επιστήμη και τα επιστημονικά στοιχεία είναι απαράλλαχτα και πολύ πιστικά. Όπως ξέρετε, εξετάστηκε το έργο του IPCC σε μία μελέτη, αλλά έγιναν και σχόλια σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο υπόθηκε ότι ο κύριος Πεσάρη θα πρέπει να είναι πρόεδρος του IPCC στην επόμενη περίοδο. Αλλά ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παρατηθεί εκτός και αν το ζητήσουν αυτό όλες οι χώρες. Άρα, ποιον υποστηρίζετε σε αυτό το θέμα για την αξιοπιστία του σώματος. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Άικαουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα δούμε... Μας είπατε τι θα γίνει το 2011 και τα τρία στοιχεία που αναφέρατε είναι πραγματικά σημαντικά. Να τονίσω όμως το εξή Μετά την αποτυχία της Κοπενχάγης και ένα χρόνο ουσιαστικά απραξίας σε διεθνές επίπεδο, καιρός είναι πια η Ευρώπη να δείξει ότι έχει την ηγεσία, αν θέλετε, στον τομέα αυτό. Και πραγματικά συμφωνώ με τον συνάδελφο Γιώργενσον που είπε ότι ε, τίθεται σε αμφισβήτηση η αξιοπιστία της Ένωσης όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για τους στόχους μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα και λέμε ότι θα βασιστούμε στο διεθνές ε, επίπεδο αυτό δεν είναι σαφές, δεν δείχνει τι θα κάνουμε εμεί στο άμεσο μέλλον. Άρα θέλουμε σαφεί νομοθετικέ προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα βασικά προβλήματα. Για παράδειγμα, οι εκπομπέ στον αυτιλιακό τομέα, το ίδιο και σε ό,τι αφορά τα αέρια Πρόκειται για μέτρα τα οποία μπορεί να αναλάβει μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτόν τον τομέα θέλουμε να είναι πιο φιλόδοξη η Επιτροπή. Και τώρα για να περάσουμε στον στόχο άνω του 20% για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου άνθρακα. Είναι σαφές ότι το Συμβούλιο αναμένει πάντα μία ανάλυση κατά κράτος μέλος. Δηλαδή λέει ότι πριν αυξήσουμε το στόχο αυτό θα θέλαμε να ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά και κοιτώντα τα απορίσματα αναφέρουν ότι αναμένεται στο Εαρινό Συμβούλιο να ξαναγίνει τέτοια συζήτηση. Άρα, σε ποιο βαθμό βασίζεστε σε ανάλυση ανακρατός μέλος και πότε θα είναι έτοιμη αυτή η ανάλυση και αφετέρου. Αν τελικά υποβάλλετε πρόταση για να υπερβούμε αυτό το στόχο του 20%, Ποιο θα είναι το νομοθετικό πλαίσιο αυτό που ορίσατε στην ανακοίνωσή σας, δηλαδή κάποια δικαιώματα εκπομπών, τι μπορείτε να μας διευκρινίσετε αν ήδη επεξεργάζεστε αυτή την πρόταση για το 2011, τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα. Ένα τελευταίο θέμα για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση που θα λάβουμε μέχρι τα τέλη του έτους είτε περάσει το θέμα για τα βιοκαύσιμα και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ βασικό γιατί αν δεν καταλήξουμε σε συγκεκριμένο συντελεστή τότε ακριβώς θα υποσκάψουμε για μία φορά ακόμα την αξιοπιστία της Ένωσης. Άρα κατά πόσο προτίθεστε να σπρώξετε αυτό το μέτρο ο Πρόεδρος. Μάλιστα, εξαντλήσατε τα τρία σας λεπτά. Ο κύριος Λίζα. έχει δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο θα ήθελα να σας ενθαρρύνω, να σας ζητήσω να προωθήσετε ένα θέμα που αναφέρατε, το στόχο για το 2030. Όντως, αυτό κάνει πολύ σχετικό το κατά πόσο θα πετύχουμε κάτι μέσω πρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα. Το να ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε μακροπρόθεσμα. Να μας πείτε δύο λόγια λοιπόν παραπάνω και να μας πείτε και δύο λόγια για το 2050 και τους στόχους που θα τεθούν εκεί πέρα. Έχουμε αύριο να ψηφίσουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος, αλλά με προβληματίζει ένα στοιχείο στο σημείο 9 του ψηφίσματος, το οποίο είναι εξαιρετικό βέβαια το ψήφισμα, αλλά αναφέρει το σημείο 9 ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να πετύχουμε το στόχο του Τη μείωσης και μέχρι το 2050 80 έως 95%. Αυτό λέει η επιστημονική κοινότητα. Αυτό θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε από τη δική σας άποψη, γιατί είναι μεγάλο το φάσμα, καταλαβαίνετε. 80% είναι λίγο, 95% είναι πολύ. Ποια είναι η άποψή σας. Και τελευταίο στοιχείο, έχετε νέα από τον τομέα της, ε, των αεροπορικών μεταφορών. Έχει, υπάρχει κάποια κίνηση σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να εξευρεθεί μία λύση ή εξακολουθεί να υπάρχει ο φραγμός των, τριών, των τρίτων κρατών που δεν θέλουν να λάβουν διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θέλουν να εφαρμόσουν τέτοιες νομοθεσίες. Ευχαριστώ. Η επόμενη μιλητρία. Tack Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή αυτή που ήταν ιδιαίτερα περιεκτική και κάλυψε κάθε θέμα. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Διατρέχουμε ένα κίνδυνο να φτάσουμε στην Κανκούν και να έχουμε σε αποσκευές μας τρεις αποτυχίες ήδη. Πρώτα απ' όλα τον προπολογισμό, το είπατε εσείς ο ίδια δεν καταφέραμε να έχουμε ένα προϋπολογισμό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις αναλήψεις υποχρεώσεων στη συνάντηση της Κοπενχάγης στη βοήθεια στο κλίμα. Δεύτερο, άλλη αποτυχία. Είναι η πρώτη ευκαιρία για να αποδείξουμε το τι πραγματικά είμαστε τεθειμένοι να κάνουμε εδώ στην κοινωνία μας για τις φιλοδεξίες μας μετά από την Κοπεχά, για το κλίμα και μετά από τις ρυθμίσεις για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα, ας πούμε, την επομπή αερίων. Και σήμερα ακόμα φαίνεται ότι δεν καταφέραμε να σεβαστούμε τις φιλοδοξίες που εσείς είχατε κύριε Επίτροπε και εμείς οι σοσιαλιστές οι δημοκράτες είχαμε αλλά και άλλες πολιτικές ομάδες όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προώθησαν ας πούμε του ΕΛΚ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και η τρίτη αποτυχία ποια είναι οι φιλοδοξίες για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος για μια μείωση της τάξης του 30%. Γνωρίζουμε ότι μεγάλα κράτη-μέλη είπαν ότι θέλουν να προχωρήσουν στο θέμα αυτό, αλλά τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη δεν είπαν τίποτα, ούτε θετικό ούτε αρνητικό και η χώρα μου, η Σουηδία, που είχε αναλάβει την Προεδρία και στην ε, στιγμή ακριβώς της συνάντησης Κοπενχάγης δεν ε, διστάζει για να προχωρήσει σε αυτό το φιλόδοξο 30%. Από ό,τι φαίνεται ο κίνδυνος είναι να φτάσουμε στην Κανκούν ε, με άδεια τα χέρια λόγω των αποτυχιών αυτών, των ελλείψεων αυτών. Για αυτό σας παρακαλώ συλλογιστείτε και πάλι. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε κάτι να κάνει το Συμβούλιο να βεστοποιηθεί πάνω σε αυτό που θέλουμε και εμείς οι πολιτικές ομάδες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε περισσότερη υποστήριξη από εσάς. Κορίν Λεπέζ. Κύριε Επίτροπε, να σας ε, ευχαριστήσω για την εισήγησή σας. Το 2011 η Επιτροπή θα μπορούσε να μας προτείνει αυτή τη μείωση του 30% γιατί με σε εκπομπές αερίων, αλλά πέρα από αυτό τώρα, σε δύο σημεία να σας απευθύνω μια ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, την άμμο με πίσα αυτό το μείγμα, αλλά παρακαλώ προσέξτε κάτι για τις προσπάθειες αύξησης εξόρυξης πετρελαίου. Εάν είχαμε μια αύξηση εξόρυξης πετρελαίου μέσω εξεδρών offshore και με τα συστήματα αυτά, τότε δεν μπορούμε που να σεβαστούμε αυτή την πολιτική μας για τη μείωση εκπομπών αερίων με, που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου. Για αυτά τα μείγματα, μου πείσας και λοιπά, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε και τι γίνεται με την εκτίμηση. Δεν έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα. Αν δεν έχουμε μια τιμή ε, των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τότε η πραγματική οικονομία δεν θα έχει καμία σχέση με την οικολογική έμπνευσή μας και προσπάθειά μας. Εντάξει, Κακόμα κάτι δεύτερο. Για τα καύσιμα και την ποιότητά τους. Η... Στην Επιτροπή έχει δοθεί μια εντολή για μια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή η 31 Δεκεμβρίου που προβλέπεται μέχρι τότε το θέμα αυτό και επειδή έχω ξεπεράσει το χρόνο μιλίας μου και ευχαριστώ τον Πρόεδρο που με καλό μεταχειρίζεται. Λοιπόν, ε, αυτό ότι αυτή η έμεση αλλαγή διαχείριση του εδάφους ε, ε, παίζει ένα ρόλο κατάλληλο γιατί αν δεν το δούμε αυτό δεν θα έχουμε μια ακριβή εικόνα όσον αφορά την οικολογική πραγματικότητα των πραγμάτων ε, για τα αγροκάψιμα. Ευχαριστώ. Επόμενος. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε, κυρία Επίτροπε, στο ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να τηρήσει μια ενιαία στάση και ξέρουμε ότι το προηγούμενο έτος το πετύχαμε αυτό, δεν είχαμε ε, ενιαία στάση ως Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους. Και να πω το εξή: εδώ μιλάμε για το ποσοστό μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα και για την ε, δυνατότητα πώληση ποσοστώσεων μετά το 2012. Τα μονομένα κράτη έχουν πολύ διαφορετική ιστορία και παρελθόν. Και φυσικά ανοίγονται και πολλές διαφορετικές ευκαιρίες σε κάθε κράτος μέλος. Η Πολωνία στο Κιώτο υποσχέθηκε 6% μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και πέτυχε το 13%. Η Ρουμανία υποσχέθηκε 8% και πέτυχε 37% και πολλές χώρες άλλες ε, ουσιαστικά πέτυχαν πολύ παραπάνω από αυτά που είχαν δεσμευθεί και πολλές χώρες είχαν θέσει ε, φιλόδοξους στόχους τους οποίους δεν πέτυχαν, συνέβη το αντίστροφο δηλαδή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε το εξής. Τα κράτη που αναφέρθηκαν και τα κράτη της Βαλτικής, η Τσεχία, η Σλοβακία, χωρίς τις χώρες αυτές οι οποίες πέτυχαν πολύ παραπάνω από τις αρχικές τους δεσμεύσεις. Χωρίς λοιπόν αυτές τις χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχε πετύχει τους στόχους που η ίδια έθεσε. Ως εκ τούτου λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορούμε να ηγηθούμε του αγώνα αυτού κατά της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος τα κράτη, αυτά που πέτυχαν ε, παραπάνω από αυτά που είχαν υποσχεθεί, θα πρέπει να τιμωρηθούν τελικά. Δεν μας επιτρέπει η Ένωση, δεν θέλει να μας επιτρέψει να πωλήσουμε τέτοιες ε, ποσοστώσεις μετά το 2012. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κοινή θέση στις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό τελικά δεν μας επιτρέπει να έχουμε κοινή θέση. Τι έχει γίνει λοιπόν τους τελευταίους μήνες για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Κρήτον Αρσένης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε θα άθελα να αφαιρθώ και εγώ σε αυτό το οποίο υπόθηκε για την ασφαλτούχο άμμο και για άλλες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ σημαντικό για τη δική μας την Επιτροπή. Μας είπατε ότι προτίθεστε να βελτιώσετε τον τρόπο με τον οποίο μελετάμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εκτίμησή του μέχρι το 2011. Θεωρώ όμω ότι θα έπρεπε να είχαμε κάτι ήδη νωρίτερα, γιατί ήδη έχουμε 12 μελέτε που μα δίνουν κάποιε εκτιμήσει για τι κλιματικέ αλλαγέ. Επίση, κάτι ακόμα, κύριε Επίτροπε. Είπατε ότι οι Κινέζοι προχωρούν γρήγορα και το εμεί χάνουμε την ανταγωνιστικότητά μα. Μήπω αυτό ακριβώ περιμένει η Κίνα προτού συμφωνήσει για μια παγκόσμια συνθήκη για το κλίμα. μήπω ακριβώ αυτή είναι η τακτική τη. Ευχαριστώ. Okay. Σα λοιπόν, um, Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για το Κανκούν. Καταρχάς, θα πρέπει να δούμε πού έχουμε σημειώσει πρόοδο μέσω της Κοπενχάγης και να περάσουν αυτά τα σημεία στις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά όλες οι συναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν τις υποσχέσεις τους, να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Διαφορετικά θεωρώ ότι το ηθικό στο Κανκούν θα είναι πολύ αρνητικό. Όλοι πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Έπειτα πρέπει να θέσουμε κάποιες φιλόδοξες ε, υποσχέσεις, κάποιους φιλόδοξους στόχους. Πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τα όσα έχουμε ξεκινήσει στις πραγματεύσεις για τα δάση, για την τεχνολογία και στο το Νοέμβριο η ομάδα του Μπάνκι Moon θα καταλήξει κάποια απορίσματα και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για την μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική ευτεκτονική Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε τα όσα λέγονται για το MRV στην ε, Συμφωνία της Κοπενχάγης και νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να εμπλουτιστεί με περισσότερες λεπτομέρειες το MRV γιατί ε, συζητήθηκε σε πάρα πολλές επίσημες και άτυπες συναντήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να σημειώσουμε πλέον πρόοδο. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία θα έλεγα. Αυτό που είναι επίση πολύ σημαντικό είναι η συμφωνία να είναι σωστά ισορροπημένη, προκειμένου να θέσω τα πράγματα με τον πιο άμεσο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς δεσμεύεται και θέλει να προχωρήσει όσο το γρηγορότερα στην, στο Κανκούν και αυτό είχε κάνει και στην Κοπενχάγη. Το σημαντικό όμω να καταφέρουμε να πετύχουμε μια μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση χωρίς τη χρηματοδότηση αυτή δεν μπορούμε να πετύχουμε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Επίσης, δεν μπορούμε να συμφωνούμε με το πρωτόκολλο, αλλά να μην κάνουμε τίποτα στον τομέα του LCA. Και εκεί θα πρέπει η στάση μας να είναι ισορροπημένη. Επίσης, για την περίοδο, τη δεύτερη περίοδο των δεσμεύσεων. Ορισμένοι αναρωτιούνται θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων για την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό στο Κανκούν. Και αυτό γιατί τα περισσότερα συμβαλόμενα μέρη συνειδητοποιούν ότι αν κάναμε κάτι τέτοιο, χωρίς να θέσουμε κανέναν όρο, καμία συνθήκη και δεν δεσμευτεί μετά ούτε η Ρωσία, ούτε η Ιαπωνία, ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, τότε στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται η δική μας η στάση να συμβάλλει καθόλου από περιβαλλοντικής πλευράς. Δεν θα μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα καθόλου. Εμείς σαφώς θέλουμε μια συμφωνία η οποία είναι νομικά δεσμευτική. Σαφώς ε, θέλουμε να προσυπογράψουμε σε πάρα πολλές δεσμεύσεις, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε εμείς κάτι τέτοιο μονόπλευρα, χωρίς να δεσμεύονται και άλλες αναπτυγμένες χώρες. Υπάρχουν κάποιοι τομείς του πρωτοκόλλου του Κιώτο ακόμα που δεν έχουν κάποια περιβαλλοντική ακαιρεότητα. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Ορισμένοι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συγγνώμη, θα μπορούσε να δεσμευθεί μέχρι το 2018. Μα αν κάναμε κάτι τέτοιο, τι θα συνέβαινε. Αυτό που θα συνέβαινε είναι το ακόλουθο δεν θα ασκούταν πλέον καμία πίεση στους Αμερικάνους προκειμένου να δεσμευτούν και αυτοί για την περίοδο μέχρι το 2018. Και το ίδιο θα ίσχυε και για άλλες χώρες. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να, είναι πάρα πολύ, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ας μην κάνουμε πολύ θετικές ε, ή πολλά υποσχόμενες δηλώσεις, χωρίς από την άλλη να φροντίζουμε να δεσμεύονται και οι άλλοι εταίροι και τα άλλα συμβαλόμενα μέρη. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τον Ιωάννης Χάνς προκειμένου να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από τα περιφερειακά διαρθρωτικά ταμεία. Είναι πολύ σημαντική ε, η συμβολή εδώ πέρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, γίνονται και διάφορες προτάσεις για να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα. Πολλά πράγματα θα μπορούσε να γίνει, να έχουμε δεσμεύσεις πλέον για τα φορτηγά. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα τα οποία θέλουμε εμεί να προωθήσουμε και στα οποία θέλουμε να εντάξουμε τη διάσταση τη κλιματική αλλαγή, αλλά περιμένω και τη συνεργασία και τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαστε ειλικρινεί. Όσο πιο συγκεκριμένε και ειδικέ προτάσει κάνετε εσεί τόσο το καλύτερο. Και προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι για το 20% πριν το 2020. και μόνο στον χώρο αυτό μπορούμε να είμαστε πιο, πιο φιλόδοξοι, δηλαδή στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι πολύ σημαντικές λοιπόν οι προτάσεις που θα βγουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω επίσης κάτι ακόμα όσον αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπα ότι δεν άλλαξε από την Κομπεχάγη και μετά, όχι. Ενδεχομένως όμως η Ευρώπη είναι αυτή που δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε στην Κοπεχάγη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, ρωτάτε, διαρωτάστε αν οι συνθήκες θα είναι οι κατάλληλες, αν θα έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλοι όροι. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι έπρεπε να πούμε ότι το ζήτημα δεν είναι να προσπίσουμε μόνο τα συμφέροντα μιας διεθνούς σύμβασης, αλλά να θέσουμε στο προσκήνιο και τα ίδια τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνει αν, για παράδειγμα, δεν προχωρήσουν οι πραγματεύσει σε διεθνέ επίπεδο. Θα μείνουμε εδώ πέρα, θα τελματώσουμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να κάνουμε τίποτα. Αν οι υπόλοιπε χώρε αποφασίσουν να μην ακολουθήσουν το δικό μα στόχο του 20%, εμεί θα παραμείνουμε σε μια κατάσταση μπλοκαρισμένη. Είναι πολύ καλό να βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι, συμφωνώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να θέτουμε στο προσκήνιο και τα δικά μα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Πιστεύω ότι θα πρέπει εμεί τουλάχιστον να είμαστε φιλόδοξοι και νομίζω ότι έχουμε συμβάλει πολύ, έχουμε κάνει τις απαραίτητες οικονομικές αξιολογήσεις εκθέσεις μας και να πρόκειται πλέον στα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση. Και όπως είπατε, ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές, έχουν υποβάλει εκθέσεις, αλλά ας το παραδεχθούμε, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν εξκαθαρίσει ακόμα τη στάση τους. Τον Οκτώβριο θα έχουμε το Συμβούλιο Υπουργών ε, Οικονομικών. Υπάρχουν όμως ακόμα πάρα πολλέ χώρες οι οποίε δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα. Ακόμα διαμορφώνουν δηλαδή τη στάση τους. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι το IPCC έχει προτείνει το στόχο του 25%. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι στο Κανκούν δεν θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τους ε, στόχους μείωσης γιατί οι Αμερικάνοι δεν έχουν ακόμα δεσμευτεί, αλλά μετά το Κανκούν θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα πολύ έντονα και αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε υποβάλει ήδη πάρα πολλά στοιχεία. Κάποιοι ρώτησαν τι κάνουμε με τα κράτη-μέλη, μα περιμένουμε κάθε κράτος μέλος αυτή τη στιγμή να αναλάβει δράση. Γίνονται, ξέρω, κάποιες συναντήσεις. Έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολλοί γενικοί διευθυντέ, πάρα πολλοί εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που προσπαθούμε εμεί να κάνουμε είναι να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώ θα υπολογιστεί το κόστο τη πολιτική μα αυτή, αλλά και πώ θα μεταφραστεί σε εθνικό κόστο για κάθε κράτο μέλο ξεχωριστά. Είναι σημαντικό το κόστος να είναι σωστά κατανομημένο και να βασίζεται σε πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας. Και αν το βάρος το μεγαλύτερο το φέρουν ορισμένα κράτη-μέλη, τότε θα πρέπει, πιστεύω, οι πολιτικές μας να συνδεθούν περισσότερο με τις δυνατότητες που μας δίνονται από τις α, δημοσιονομικές προοπτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον κοινωτικό προπολογισμό. Ο Chris Davis αναφέρθηκε στην, ηγεσία, την, Αμερικανική, την αμερικανικής ηγεσία, συμφωνώ και θα έλεγα ότι αυτό κάνει και πάρα πολλές άλλες χώρες να κρύβονται πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αναφέραμε αυτό σε όλες τις δημαρείς επαφές που είχαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι ότι στις ενδιάμεσες αυτές εκλογές που γίνονται εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα το πάρα πολύ σημαντικό Καταγράφουμε πάντως την κατάσταση και συμφωνώ μαζί σας ότι ε, η απουσία αυτή η πρωτοβουλία των ΗΠΑ καταστά την όλη διαδικασία πολύ πιο δύσκολη. Καταλαβαίνετε επίση ότι είναι πολύ σημαντικό να δεσμευτεί νομοθετικά επίση η Αμερική, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από το Κανκούν. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ φιλόδοξο όσον αφορά του στόχου που έχουμε θέσει για τη μείωση των εκπομπών και εμείς έχουμε βασιστεί στην δική σας συμβολή και να αναφερθώ επίσης λίγο και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με την καινοτομία τις νέες τεχνολογίες όσον αφορά τα γιοταχή. Αυτή τη στιγμή το ότι καταφέρνουν πάρα πολλές εταιρείες να παρουσιάζουν νέα καινοτόμα αυτοκίνητα οφείλεται στο ότι εμείς πριν από μερικά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλαμε νέους κανονισμούς και οδηγίες οι οποίες οδήγησαν την αυτοκινητοβιομηχανία στο να κάνει τέτοιες προτάσεις. Εφόσον η αυτοκινητοβιομηχανία αυτή τη στιγμή δέχεται τι προτάσει μα και κατασκευάζει νέα οικολογικά αυτοκίνητα, μήπως θα έπρεπε να πείσουμε και την αυτοκινητοβιομηχανία, με συγχωρείτε, αλλά και του άλλου τομεί, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά έχει δίκαιο όταν προτείνει κάποιου φιλόδοξου καινοτόμους στόχους και στη συνέχεια οι επικληματικοί κλάδοι ακολουθούν, γιατί θα θυμάστε ότι η αυτοκινητομηχανία έχει αντιδράσει αρνητικά στην αρχή. Επίση, να αφαιρθώ λίγο στο IPCC. Εμεί δεν έχουμε επίσημο ρόλο σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ένωση στην διοικητική διάρθρωση του IPCC. Το IPCC, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματο, είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίσει για την ηγεσία τη να απαντήσω και στον κύριο Γιάκομψεν για την ανάλυση των κρατών μελών. Μέχρι στιγμής οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, μάλλον οι αρμόδιοι υπουργοί από κάθε χώρα, έχουν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και η Δανία επίσης πριν από μια εβδομάδα δεσμεύτηκε για τους στόχους μείωσης εκπομπών δικτύου του άνθρακα είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν όλοι και περισσότερε χώρε που επιθυμούν φιλόδοξου στόχου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ρωτήσατε πώ θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο του 20%. Στα έγγραφά μα περιγράφουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φτάσουμε στο στόχο αυτό. ETS, νέα μέτρα για τη γεωργία, χρησιμοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, όλα αυτά είναι χρήσιμα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο Πίτερ Λίζε δεν ξέρω αν κατάλαβε πολύ καλά την ερώτησή σας. Αναφερθήκατε στο, στο 80%. Κοιτάξτε, ξέρω ότι σε πάρα πολλές διεθνείς διαπραγματεύσεις αναφερόμαστε απλώς σε ένα 5%. Και καταλαβαίνετε ότι στις διεθνείς διαπραγματεύσεις έχουμε και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Αν εμεί ω αναπτυγμένο κόσμος δεν θέσουμε τους πιο φιλόδοξους στόχου για το 2050, τότε οι αναπτυσσόμενε χώρες φοβούνται ότι το δικό τους μερίδιο εκπομπών δεξιού του άνθρακα θα είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Και ο λόγος που δεν καταφέραμε να, πετύχουμε έναν παγκόσμιο στόχο 50% στην Κοπενχάγη έχει να κάνει με τους φόβους που τρέφουν αυτή τη στιγμή η Ινδία, Κίνα και άλλες χώρες ότι θα έχουν ένα πολύ μειωμένο περιθώριο εκπομπών δεξιού του άνθρακα. Αν λοιπόν να θέσουμε στόχο το 80% θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και δεν θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε στον μακροπρόθεσμο στόχο του 50%. Αν υπάρχουν ε, αλλαγές στον τομέα της αεροναυτιλίας, όχι. Είδα ένα νέο σχέδιο κειμένου το οποίο διαπραγματευόμαστε σήμερα. Σίγουρα οι φιλοδοξίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Όσοι συνεργάζεστε για τον τομέα αυτό θα γνωρίσω ότι στο τέλος της εβδομάδας όταν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του, ΙΚΑΟ θα γνωρίζουμε αν έχουμε πετύχει κάποια πρόοδο ή αν βρισκόμαστε στην κατάσταση που είχαμε, που πριν από μερικά χρόνια. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολε οι πραγματεύσει στον τομέα αυτό και υπάρχουν πολλά συμβαλόμενα μέρη τα οποία διαφωνούν με τη δική μα τοποθέτηση. Η κυρία Ουλσκούκα αναφέρθηκε σε κάποια κενά που υπάρχουν στον προπολογισμό. Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι προσπαθούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Η Βελγική Προεδρία θα προσπαθήσει σε πρώτη ανάγνωση να διευθετήσει το ζήτημα αυτό και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε το συντομότερο δυνατό να κάνουμε κάποιες φιλόδοξες προτάσεις. Και όσον αφορά το 7% αναφέρθηκε και σε αυτό, μας είπατε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου το Συμβούλιο να κάνει αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να κάνει Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε να του παρουσιάσουμε κάποια καλά κέρια επιχειρήματα, να τους δώσουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία, επιστημονικά δεδομένα και να πρόκειται πλέον σε εμά να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να τα πείσουμε ότι ε, ε στη τελευταία ανάλυση η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων για την κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε μια καλύτερη οικονομία και σε ένα καλύτερο επίπεδο ανταγωνιστικότητα. Πιστεύω ότι ε, ο κίνδυνος της ε, διαρροής ε, στο σύστημα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι ένας υφιστάμενος κίνδυνος, αλλά ενδεχομένως να καταφέρουμε, μάλλον να καταλήξουμε σε απώλεια θέσεων εργασίας, αν δεν είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να κρατήσουμε την κατάλληλη ισορροπία, λαμβάνοντας υπόψη μας και τον κίνδυνο διαρροής. Η κυρία Λαπάζ αναφέρθηκε στη στάση που έχουν πολλοί βουλευτές στα πλαίσια της Επιτροπής σας. Δεν συμφωνώ όμω με αυτό το οποίο είπατε ότι δεν έχει γίνει καμία αναφορά, ότι δεν ξέρετε πού θα καταλήξουμε ακόμα. Εγώ σε πάρα πολλές ε, γραπτές απαντήσεις που έχω δώσει στην επίσημη ανταλλαγή απόψεων, αυτό που λέω είναι ότι κάνουμε μία ανάλυση για την ασφαλτούχο άμμο, ακριβώς όπως κάναμε και στο παρελθόν. Όταν ε, ήρθα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνειδητοποίησα ότι ο τομέας αυτός της ασφαλτούχου άμμου δεν ε, αξιολογεί το όπως άλλοι τομείς. Πίεσα λοιπόν προκειμένου να καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε την ίδια μεθοδολογία και στην ασφαλτούχο άμμο όπως χρησιμοποιούμε σε άλλους τομείς. Γι' αυτό το λόγο ζήτησα από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν τα τέλη του έτους να υποβάλουν μία ανάλυση προκειμένου να ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε. Ήδη όμως από τώρα έχουμε στείλει το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη αξιολόγηση, μια συγκεκριμένη αποτίμηση της αξίας της ασφαλτούχου άμμου. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό οι αρμόδιοι και ότι θα έχουμε σύντομα μία, μία συγκεκριμένη τοποθέτηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Υπάρχουν κάποιε διαπραγματεύσει οι οποίε θα ολοκληρωθούν στο τέλη και εμεί ασκούμε πίεση για να ολοκληρωθούν το στομότερο δυνατό. Τέλο, με ρωτήσατε για το AAU. Γίνεται μια πολύ σημαντική και δύσκολη συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Έχουμε δισεκατομμύρια τόνους θερμού αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσό υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ακόμα στην ε, Ρωσία. Το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη στις πρωτοβουλίες μας και είναι πολύ σημαντικές συζητήσεις που πρέπει να γίνουν για αυτό το ζήτημα. Ξέρω ότι για πολλά κράτη-μέλη το ζήτημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Η συζήτηση δεν διεξάγεται εύκολα τα πράγματα όμως θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν καταφέρουμε να λύσουμε αυτό το αδύναμο σημείο της, ε, του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι διακινδυνεύουμε να έχουμε 8 δισεκατομμύρια τόνους θερμού αέρα, hot air, τα οποία θα έρθουν από τη Ρωσία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι Προτού είναι πολύ αργά, θα πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Ελπίζω να έχετε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να έχετε χρόνο και πέρα από τι 4.30, γιατί αλλιώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ε, ε, διαπραγματεύσεις μας, ε, τις συζητήσεις μας. Δύο λεπτά για τους υπόλοιπου ομιλητές, γιατί δάλλως δεν θα, δεν θα προλάβουμε. Η κυρία Χάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Επίτροπε, καλύψατε πάρα πολλά θέματα. Θα ήθελα ωστόσο να σας ε, θέσω άλλα δύο ζητήματα. Καταρχάς, ε, η ενεργειακή σήμανση των επιβατηγών αυτοκινήτων. Μια χαμένη ευκαιρία σε ό,τι αφορά την νομοθεσία. Μιλήσατε για τα αυτοκίνητα και είπατε ότι αποτελούν ένα καλό παράδειγμα σε ό,τι αφορά την, ε, τα πρότυπα για την αυτοκινητοβιομηχανία. Γιατί δεν χρησιμοποίησαμε όμως την σήμανση ενεργειακής αποδοτικότητας για τα α, επιβατικά αυτοκίνητα. Κατά δεύτερον, αναφερθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για την περιβαλλοντική αικαιρότητα και τις ε, Ένωσης και πέρα από την Ένωση. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια παραπάνω. Ποια είναι η δική σας άποψη. Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά την... Ε, ποιος θα πρέπει να είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρήση των γεών. Ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστούμε και την ε, Επίτροπο για την ειλικρινή της ε, στάση. Είναι τεράστια η ευθύνη σας, ίσως και μεγαλύτερη από αυτή που θεωρείτε εσείς, γιατί βρισκόμαστε πριν από το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στην Ολλανδία και ουσιαστικά διαγράφησαν όλες οι δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, εξαρτώνται τελείως από εμάς. Σας παρακαλώ λοιπόν να συνεχίσετε την καλή σας δουλειά για τον λαό της Ολλανδίας. Μια συγκεκριμένη ερώτηση να σας κάνω. Μιλήσατε για την εξουδετερώση, αν θέλετε, ε, του προπολογισμού σε ό,τι αφορά το κλίμα. Έχω υποβάλει πολλά ερωτήματα στο παρελθόν και μου έχουν απαντήσει οι συνάδελφοί σα από την Επιτροπή, αλλά δεν με έχουν ικανοποιήσει οι απαντήσει αυτέ τα επίπεδα ανακράτο μέλο. Να σα ρωτήσω το εξή. Έχετε κάποια συγκεκριμένη ατζέντα για την αντιμετώπιση του θέματο. Ο Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ ε, Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Συνεχίζουν οι αμφιβολίες μου. Εάν δεν υποβληθεί μια πολιτική πρόταση που να λαμβάνει υπόψη της, τις δηλώσεις του Μπαλί, τότε δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και κάτι να πω ακόμα και να επιμείνω απαιτείται ένα σύστημα ανταλλαγής εκπομπών ε, που να είναι πιο απλό και πιο γενικό. Και έτσι ουσιαστικά να φτάσουμε σε μια δικαιοσύνη κλιματική στην οποία αναφέρθηκε ήδη το Κοινοβούλιο και μάλιστα πρόσφατα. Κάτι ακόμα να τονίσω. Κατά την άποψή μου, η συζήτηση για το 20 ή 30% για το 2020 δεν τίθεται πλέον το θέμα αυτό. Αποδείχτηκε σε πολλές πλευρές του κόσμου ότι το 2050 θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό εάν δεν χρησιμοποιούμε πια καθόλου άνθρακα. Α, λοιπόν, εμείς, ειδικά εμείς θα πρέπει να το κάνουμε. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από κρίση. Αυτό που απαιτείται είναι επένδυση ιδιαίτερη στο μέλλον μας. Και αυτό μπορεί να γίνει κατά την άποψή μου. Και να σας πω ότι συμμετέχω στην ομάδα εργασίας ε, για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές που συνέστησε η Επιτροπή. Και θα πρέπει στη βάση αυτή να το σκεφτούμε για μια προσαρμογή που να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο του συστήματος και όχι κατακαιρματισμένα όπως βλέπω να διατρέχουμε τον κίνδυνο. Ευχαριστώ Φλόρεντς. Ο κύριο Φλόρεν, θα ήθελα να σα ρωτήσω και άλλα πράγματα για την αυτοκινητοβιομηχανία. Τέλο πάντων, να πω το εξή. Μ' ανησυχεί λίγο το γεγονό ότι πολλοί εξημών λένε ότι θα πρέπει να μιλάμε με μία φωνή στο Κανκούν. Κοιτώντα όμω τι τροπολογίε που θα ψηφίσουμε αύριο, πρέπει να πω ότι ούτε εμεί είμαστε σύμφωνοι. Άρα, τι ακούγεται στο Συμβούλιο συγκεκριμένα ακούγονται φωνές από χώρες που λένε ότι δεν θέλουν να μιλάμε με μία φωνή. Να μιλάμε με πιο πολλές φωνές, δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχετε και επαφές με τον ΟΗΕ. Ποια είναι τα μηνύματα που ακούτε από εκεί. Σε θέματα ενεργειακής αποπτικότητας ε, φαντάζομαι ότι θα είναι πιο ανοιχτέ οι απόψει που ακούγονται. Δύο-τρει προτάσει, αν θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμπάνιο. Euh, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πρώτη παρέμβαση περίμενα τις απαντήσει σας για να, ξεκι... για να αλλάξω τα πράγματα εδώ. Ε, αυτό περίμενα. Αλλά δεν θα τα αλλάξω γιατί αυτό που κατάλαβα είναι ότι υπάρχει κάτι, μια καταπίεση, εντάξει μιλάτε με όμορφα λόγια, μιλάτε για φιλοδοξία και στη συνέχεια περιμένουμε μια συγκεκριμενοποίηση αυτή τη φιλοδοξία. Μιλάμε για τα κράτη-μέλη, μιλήσατε για κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη. 20 φορέ το είπατε στην εισήγησή σα στα λόγια σα. Καταλαβαίνουμε, όπω λοιπόν, όπως είπα και ο Φλόρενς, ότι αποδίδεται σημασία στο βάρο τη σημασία αυτών των κρατών αλλά και την αδυναμία την πλήρη, αυτό το δεύτερο μέρος που μου φάνηκε ιδιαίτερα σημαντικό στα λόγια σας, αυτή την αδυναμία, την ανεκανότητα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης απέναντι στα κράτη-μέλη. Και σημαντικό ιδιαίτερα μου φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρα από τη δική σας ε, ε, πλευρά και δεν άκουσα από τον πρόεδρο Μπαρόζο όταν χάραξε τους κύριους άξονες πολιτικής τους πριν από λίγους μήνες να μας μιλάει για φιλοδοξία πραγματική ευρωπαϊκής, ευρωπαϊκού χαρακτήρα κατά της υπεθέρμας του πλανήτη και απέναντι όμως και στην, ε, στα οικονομικά θέματα που γνωρίζουμε και που είναι από τα σημεία κλειδιά. Και κάτι ακόμα, ο ακρογωνίος λίθος της Κοπενχάγης ε, πριν από την Κανκούν ε, να μπορεί να μεταφραστεί κάπως συγκεκριμένα αυτό το πράσινο, τα πράσινα κονδύλια, ο φόρος για τις διάφορες συναλλαγές. Δεν είδαμε τίποτα ε, μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το και στις νότιες χώρες έχουμε ενέργειες για ε, νεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τι θέλει για να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, πέρα από την Κίνα που θα επιθυμούσε ίσως μια εταιρική σχέση. Θόδωρος Κυλακάκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Χάρηκα ιδιαίτερα με αυτό που είπατε για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Έχω την αίσθηση ότι πολύ συζητάμε αλλά δεν κάνουμε, δεν πράττουμε αρκετά. Είδαμε την πολιτική μας για τους υποχρεωτικούς στόχους ως προς την εκπομπή ε, του άνθρακα στο Κιώτο. Ουσιαστικά κανείς δεν θέλει να δοθεί μια παράταση, μια δεύτερη περίοδος. Η και η Κίνα δεν συμμετέχουν. Γιατί να μην κοιτάξουμε λοιπόν να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους, πολύ πιο φιλόδοξους στόχους σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ως εναλλακτική, αν θέλετε, η συμπληρωματική λύση σε ό,τι αφορά την ε, αναγκαστική μείωση, την δεσμευτική μείωση των εκπομπών. Αυτό ίσως να είναι πιο αποδεκτό από τους εκλογείς μας και ενδεχομένως να τους οδηγήσει να μας οδηγήσει σε μια πολιτική για την αλλαγή του κλίματος σε ένα τομέα όπου, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν βλέπουμε σήμερα μεγάλη πρόοδο. Κάτι άλλο που ήθελα να θίξω. Θέματα προσαρμογής. Μιλήσατε για τις προτεραιότητες και το σχετικό budget, τη σχετική χρηματοδότηση. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν υπάρχει επαρκής έρευνα σε σχέση με το τι θα συμβεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με την αλλαγή του κλίματος στην Λευκή Βίβλο συμπεριλήφθησαν όσα είπε και η IPCC, ο Διεθνής Οργανισμός, η Κυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος πριν από πέντε χρόνια. Έκτοτε όμως προέκυψαν πολλά θέματα για τα... Ε, προέκυψαν πολλά προβλήματα σε σχέση με στοιχεία που είχαν ερευνηθεί για τα Ιμαλάια, προέκυψαν σφάλματα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει πιο πολύ έρευνα προτού καταρτιστεί ε, πολιτική προσαρμογή στην Ένωση. Ο κύριος Πέτερλε. Ε, θα ήθελα να πω το εξής. δεν έχουμε από τα τρία όργανα της Επιτροπής ε, έγγραφα που να μην έχουμε τα σημεία κλειδιά, τις λέξεις κλειδιά που να μην αναφέρονται ακριβώς στρατηγική, ολοκληρωμένη λύση, η φόρος ανάπτυξη. Και αρκετοί επίτροποι μίλησαν για υποδειγματικές αλλαγές οι οποίες απαιτούνται να δώσουν το παράδειγμα μετά από την πρώτη χρονιά των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι γίνεται υγεία, μεταφόρες, γεωργία, ενέργεια, περιβάλλον, πώς συνδυάζονται όλα αυτά, τι δόθηκε σαν υπέροχο παράδειγμα και στην ε, συνεργασία αυτών των γενικών επίσης διευθύνσεων τι γίνεται που ασχολούνται με αυτούς τους τομείς για τα πράγματα εξαρτώνται από τις σχέσεις τους διάφορους τομείς από εκεί εξαρτάται και η επιτυχία των κοινών μας προσπαθειών μπορείτε να μας πείτε κάτι ακόμα με ποιο τρόπο ε, επεξεργάζεστε αυτά που ε, λέγατε παλιά ότι θα τα υπέροχα παραδείγματα Ευχαριστώ, ευχαριστούμε την ε, Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή. Δύο σχόλια. Να τονίσω ότι έχει σημασία στην περίπτωση αυτή, στη Κανκούν, να μπορέσουμε να εκφράσουμε μία και μόνο ενία φωνή και πέρα από την Κοπενχάγη Τώρα τι γίνεται από την Κοπεχάγη, από τη Δανία, από τη Γερμανία που έρχονται τα πράγματα από τη στιγμή που δεν είχαμε μία φωνή. Χρειάζεται μία, μία φωνή. Κάτι ακόμα. Σίγουρα υπάρχουν και εθνικά συμφέροντα. Οι Επίτροπος, ας πούμε, ο Ισπανός και ο Γερμανός Επίτροπος, ίσως ε, υπερασπίζονται τις εθνικές τους παραγωγές όπως τον άνθρακα. Τι γίνεται, τι γίνεται με τους επιτρόπους και για το 2014 που είπαν ότι σε παρόμοιες δραστηριότητες θα κοπούν οι επιδοτήσεις στα κονδύλια. Στην Ισπανία όμως θα διατηρηθεί η βοήθεια α πούμε στην ανθρακοριχεία. Αυτό είναι καταστροφή ε, και είναι και ένα μήνυμα αρνητικότατο που ε, δίδουμε και στους υπόλοιπους και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τι γίνεται, θέλουν ακόμα να δίνουν κρατικές επιδοτήσεις σε αυτόν τον τομέα εσείς κύριε Επίτροπε θα πρέπει να βοηθήσετε να υπάρχει συνοχή ανάμεσα σε όλους τους επιτρόπους απέναντι σε παρόμοια θέματα γιατί δεν θέλω να βλέπω επιτρόπους που είναι ε, υπέρ μοντέλων ανάπτυξης και παραγωγών. Εδώ ε, ίσως θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση από το Κοινοβούλιο ούτε και στις χώρες αυτές, στην Ισπανία και στη Γερμανία. Αλλά αυτό με τις δύο χώρες, ε, μήπως μπορείτε να απαντήσετε κάτι. Τι γίνεται, γιατί είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πάλι καλά που η Δανία έχει ολική ενέργεια και δεν χρειάζεται τον άνθρακα. Ευχαριστώ. Η Σάτουχα μίλησε για την ε, οδηγία για την επισήμανση των οχημάτων. Θα ήθελα να ρωτήσω, θα το εξετάσετε αυτό φέτος, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Στο ETS, το σχέδιο εμπορίας ρήπων, συμπεριλάβαμε την ε, αεροναυτιλία και ζητήσαμε να συμπεριληφθεί και η ναυτιλία. Πού, πώς πάει αυτή η πρόταση, τι έχει γίνει. Και τέλος αναφερθήκατε σε ένα στόχο για το 2030 για το κλίμα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Thank you, Chairman. ευχαριστώ, ευχαριστώ Λίντα που αναφέρθηκες σε αυτά τα καύσιμα. Το ίδιο ισχύει και για την αεροναυτιλία. Μιλήσατε για τη μία φωνή που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει. Πρότεινα ήδη στην ακρόασή σας να υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος, για τις συμφωνίες, τις σχετικές, στο ευρύτερο πλαίσιο. Μπορείτε να το προτείνεται αυτό, μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης για τέτοια θέματα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της αποδοτικότητας των πόρων για την μείωση των εκπομπών μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, τη βιώσιμη των αποβλήτων. Ξέρουμε ότι πολλά μπορούμε να πετύχουμε έτσι. Ξέρουμε ότι η αποδοτικότητα των πόρων είναι, αν θέλετε, το χαρακτηριστικό με το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Κακούν πριν ε, γίνει και η πραγματική, αν θέλετε, σύνοδος για το κλίμα το 2012. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Και έχω και εγώ δύο παρατηρήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Τα benchmarks τα οποία αναφέρθηκαν. Δεν ακούσαμε ωστόσο τίποτα για το CDM και ξέρουμε ότι επικρατούν μεγάλα προβλήματα στο θέμα αυτό. Δύο λόγια, αν θέλετε. Άκουσα τι είπατε για μια δεύτερη περίοδο ε, δεσμεύσεων μετά το Κιώτο, Κιώτο 2. Ουσιαστικά δεν θα έχει δυσκολίες η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τέτοιες ευθύνες. Για το 2020 έχουμε νομοθεσία και τα περιλαμβάνει ουσιαστικά όλα. Και ακόμα και αν θα πρέπει να δεσμευτούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, αν δεν το κάνουμε, Ευτύφεται πάλι θέμα, το θέμα της κότης και του αυγού. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε εμείς τίποτα, επειδή δεν κάνουν και οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι αν θα υπήρχε μια δεύτερη περίοδος του Κιώτα θα ήταν σε καλή θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπόλοιποι θα ήταν υποπίεση για να κάνουν παραπάνω από αυτά που έχουν πετύχει. Τρίτο ερώτημα τεχνικής φύσεως. Αν θα αποστείλει αντιπροσωπεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Κανκούν, 15 άτομα. Ξέρετε ότι είναι μεγάλη δέσμευση και θέλουν πολλοί άλλοι συνάδελφοι να συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία αυτή. Πώς μπορούν να διαπιστευθούν οι συνάδελφοι αυτοί. Δεν θα έχει τόσο κρύο όπως στην Κοπενχάγη αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι ευρωβουλευτές στις αίθουσες που θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ε, να απαντήσω σε αυτούς που έθεσαν μια ερώτηση για τη σήμανση των ε, επιβατικών οχημάτων. Ξέρω ότι το ζήτημα αυτό έχει διαρκέσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί τώρα να δει τι ακριβώς θα κάνει είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε και πράγματα που μπορούν να καταλάβουν οι καταναλωτές και που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές. Καταλαβαίνω ότι δίστανται απόψη για το ζήτημα αυτό, πάντως το συζητάμε και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να αναλαμβάνουμε και πρωτοβουλίες πιο κοντά στους πολίτες. Όσον αφορά τώρα το LULUCF, τη χρήση της γης, την αλλαγή της χρήσης της γης και τις δασακομικές δραστηριότητες, νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί μία λύση στο πρόγραμμα καταγραφής που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπως η Φιλανδία που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να βρούμε μία και μοναδική ευρωπαϊκή τοποθέτηση για το ζήτημα αυτό και να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μία συμβιβαστική λύση, προκειμένου να είναι συνεκτική και συνεπή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλάμε με μία φωνή στις διεθνείς διαπραγματεύσει. Συζητά λοιπόν το ζήτημα αυτό με τα κράτη-μέλη προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε ε, ένα έτος αναφοράς κοινό για όλους. Αναφερθήκατε επίσης και σε επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές για τις επιδοτήσεις του άνθρακα, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και αυτό μπορώ να σας πω ότι έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, τις, για τους μη κερδοσκοπικούς ε, οργανισμούς ε, εξόρυξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα πρέπει να μειωθούν τα κονδύλια και είναι πολύ σημαντικό να λήξουν τα κονδύλια αυτά στα πλαίσια της υφιστάμενης εντολής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή 1η Οκτωβρίου του 2014, να μην περάσουν τα κονδύλια αυτά στην εντολή μιας νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει εκ νέου να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Αυτό είναι το πιο λογικό, αν θέλετε, από περιβαλλοντικής και οικονομικής πλευράς. Και νομίζω έπειτα ότι υπάρχει και το άλλο ζήτημα των ad hoc εθνικών επιδοτήσεων. Πάντως, και αυτές θα πρέπει να διευθετηθούν μέχρι το 2014. Από περιβαλλοντικής κλιματικής πλευράς οι επιδοτήσεις αυτές θα λήξουν μέχρι το 2014. Αυτή είναι η στάση μας. Ξέρω, διαβάζω και εγώ τις εφημερίδες, ξέρω ότι ε, το ζήτημα είναι αρκετά διαφιλονικούμενο σε διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω πως αισθάνονται ορισμένε χώρες για τα ορυχεία. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι ε, Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη, για παράδειγμα ένα, το οποίο δίνει 50.000 ευρώ ετησίως αναθέσει εργασίας όσον αφορά την απασχόληση στα ορυχεία. Καταλαβαίνετε πόσα πολλά και σημαντικά πράγματα μπορεί να κάνει μια χώρα στα πλαίσια της οικονομίας της αν χρησιμοποιήσει διαφορετικά το πολύ σημαντικό αυτό ποσό θα πρέπει σαφώ να μειώσουμε και τη χρήση των ρηκτών καυσίμων, αλλά δεν φτάνει να το κάνουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ μπορούμε να πετύχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα και στην Οδυσσία και σε άλλε συναπτυσσόμενε χώρε. Και αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει. Το ζήτημα πάντω είναι πολύ σημαντικό. Απαντώντας τον κύριο Πρόντι, καταλαβαίνω τα όσα είπατε για το 2015 και το 0% για το πόσο είναι δύσκολος ο στόχος αυτός, πόσο είναι δύσκολος για ορισμένα κράτη-μέλη. Άκουσα τις απόψει σας και του κύριου Φλόρενς ο οποίος αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να μιλάμε με μία ενιαία φωνή. Ο κύριος Φλόρενς έχει φύγει από την αίθουσα, πάντως πρέπει να πω ότι συμφωνώ αν δούμε τις δικές σας τροπολογίες και τις συζητήσεις που γίνονται στα κράτη-μέλη, να όντως υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες επί των οποίων ενδεχομένω να μην συμφωνούμε 100%. Ωστόσο, πιστεύω ότι όταν πηγαίνουμε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είμαστε αρκετά πειθαρχημένοι προκειμένου να αφήνουμε κατά μέρος αυτές τις μικροδιαφωνίες μας και να καταφέρνουμε να μιλάμε με μία ενιαία φωνή, σύσσωμα. Διαφορετικά θα καταλήξουμε στην κατάσταση που είδαμε μέχρι ενός βαθμού τουλάχιστον στην Κοπενχάγη. Στον κύριο Πανιούν να πω ότι αναφερθήκατε στο ζήτημα της παρακολούθησης του follow-up που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η στάση μας είναι αδύναμη. Εδώ και 8 μήνες ε, έχει αναλάβει τις εργασίες της η εφιστάμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που έχω εγώ να σας πω είναι ότι προσπαθούμε να προωθήσουμε όσο είναι το περισσότερο τους στόχους του 2030, του 2050. Συνεχίζουμε επί του έργου που είχε γίνει από την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασχολούμεθα με το ζήτημα της ε, φορολόγησης. Θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό σύστημα φορολόγησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε κανείς να συζητήσει περισσότερο για το ζήτημα των μεταφορών, το ζήτημα του προπολογισμού, για το ζήτημα του mainstreaming. Είναι σημαντικό να συντοπίσουμε ότι προσπαθούμε εμείς να αγγίξουμε όλα όλες τις σημαντικότερες πτυχές του ζητήματος των κλιματικών αλλαγών. Όλους τους επιμέρους αυτούς τομείς μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ο κύριος Κυλακάκης αναφέρθηκε στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Όπως γνωρίζετε αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του κύριου Ότιγκερ. Το 2011 ο αρμόδιος επίτροπος θα παρουσιάσει μια στρατηγική για το ζήτημα αυτό και είναι πολύ σημαντική βέβαια να δούμε και ποια θα είναι η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν έχουμε καταβάλει αρκετές προσπάθειες για την έρευνα. Σαφώς Υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί όπω η έρευνα και η καινοτομία που ω μια Ευρωπαϊκή Ένωση 27 κρατών μελών θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Συμφωνώ λοιπόν ότι η ενεργειακή υποδομή, οι υποδομέ που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερη καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να σε απασχολήσει. Η προσαρμογή επίση είναι ένα ζήτημα για το οποίο γίνανε συστάσει από τη Λευκή Βίβλο την περσινή Προσπαθούμε τώρα να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγης αυτούς, τους, ε, αυτές τις 30 συστάσεις για να δούμε αν καταφέρουμε τελικά να συμμορφωθούμε με αυτές. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Πέτερλε ότι θα πρέπει να συγκεράσουμε όλες αυτές τις κοινωτικές πρωτοβουλίες Απάντησα σε κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Λίντα Μακέβαν αναφερθήκατε επίσης στον ναυτιλιακό τομέα πέρα από τη σήμαση των οχημάτων. Δυστυχώς στον ναυτιλιακό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν γίνονται σπουδαία πράγματα. Γι' αυτό το λόγο ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή είπανε ότι αν δεν υπάρξει κινητικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να δούμε τουλάχιστον τι πρέπει να κάνουμε σε περιφερειακό επίπεδο. Το γνωρίζουμε αυτό και αποτελεί μέρος του προγραμματό μας. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον τομέα αυτό και οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αυτό που έγινε στον IMO την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς το ότι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι είναι προς το δικό του συμφέρον να καταλήξουν σε μία απόφαση. Από την άλλη βέβαια καταλαβαίνω ότι η ε, θέση τους είναι πολύ δύσκολη, είναι εξίσου δύσκολη με τη δική μας θέση στις διεθνεί διαπραγματεύσεις. Αυτό το οποίο λέμε εμείς ε, προς όλους αυτούς τους κλάδους είναι ότι θα εμείνουμε στις θέση μας, ότι έχουμε προσχεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ότι αν δεν υπάρχει πρόοδο σε διεθνές επίπεδο, τότε εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάτι μόνοι μας, όπως κάνουμε και για την αεροναυτιλία. Για το 2030 δεν υπάρχουν σπουδαία πράγματα που θα σας πω τώρα. Όσον αφορά όμως τους στόχους μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα 2050, δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στο σημείο κίνηση του 2020, αλλά να αναφερόμαστε και στο διάμεσο διάστημα του 2030. Δηλαδή να καταφέρουμε να θέσουμε και για το 2030 στόχους. Οι Αμερικάνοι ήδη το κάνουν αυτό στη δική τους παρέμβαση συμμετοχή στην συνδιάσκεψη της Κοπενχάγης. Επομένω, έχουμε θέλει ένα σημείο αναφοράς. όσον αφορά την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το πώς μιλάμε, αν μιλάμε με μία ενιαία φωνή. Το θέμα δεν είναι ποιος μας εκπροσωπεί, ποιος μιλάει εκ μέρους μας. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να αυτοπιθαρχηθούμε προκειμένου και τα 27 κράτη-μέλη να αποδεχθούν ότι το μήνυμα θα πρέπει να είναι κοινό, το μήνυμα θα πρέπει να είναι ενιαίο. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα θεωρώ. και η στάση μας θα πρέπει να αναφτεί και στο Κανκούν. Όσον αφορά τώρα την αποδοτικότητα των πόρων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το ζήτημα αυτό και θέλουμε και τη δική σας συνεργασία. Επίσης, ε, έχει απασχολήσει το ζήτημα αυτό και τον πάνελ της παγκόσμιας βιωσιμότητας, του οποίου ηγείται ο Μπαν Κιμούν Και πρόσφατα σε επαφές που είχαμε με το πάνελ αυτό προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια καλύτερη αποδοτικότητα των πόρων. Αυτή είναι λοιπόν η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε το πάνελ αυτό να καταλήξει κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις που θα οδηγήσουν σε ενεργειακή αποδικότητα, συγκεκριμένα παρεμβατικά μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να μπουν και στην διαδικασία, στην στρατηγική για το 2020. Τέλος, να απαντήσω και στον πρόεδρο για το CDM. Έχετε δίκιο, προσπαθούμε να κινητοποιηθούμε και στα πλαίσια του CDM. Ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις και επαφές με την Κίνα όσον αφορά τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης. Θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό, ότι έχουμε αναλάβει από κοινού κάποιες πρωτοβουλίες πρότεινα στον Υπουργό τον Κινέζο μέχρι τα τέλη Απριλίου να έρθουμε σε επαφή, μα δέχτηκε την πρότασή μας αυτή και νομίζω ότι χρησιμοποιώντας τις τομεακές αυτές συμφωνίες για την αγορά θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Είχαμε μια τέτοια επαφή ήδη τον Ιούλιο και θα έχουμε εκ νέου μια τέτοια επαφή τους επόμενους μήνες. Θέλουμε να καταφέρουμε να έχουμε ένα καλύτερο πρόγραμμα εργασίας, μια καλύτερη διάρθρωση της εργασίας μας για το CDM και να γίνει το CDM το δυνατόν λιγότερο γραφειοκρατικό προκειμένου να συμμετέχουν και περισσότερα κράτη-μέλη. Και θα μας απασχολήσει αυτό και στα πλαίσια του Κανκούν. Και εν τέλει ναι, Όντως οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελαν όντως να βοηθήσουν την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κανκούν. Σαφώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε το ζήτημα της διαπίστευσης των Ευρωβουλευτών. Ξέρετε ότι είμαστε σε επαφές κύριε Πρόεδρε για να βελτιώσουμε και το ζήτημα αυτό. Πολλές φορές σε επαφές μας υπάρχουν ε, θέματα τα οποία δεν μπορούμε άμεσα εμείς να αντιμετωπίσουμε, ξεφεύγουν κάπως των δικών μας ε, αρμοδιοτήτων. Θεωρώ πάντως ότι μέσω της δικής μας συμμετοχής μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερα και την πιο συντονισμένη δράση Μπαρόσο και Μπούζεκ. Εν τέλει να σας πω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στο Κιάντζιν της Κίνας, θα είναι δύσκολα και στο Κανκούν. Ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι σκέφτονται ότι αν δεν τα καταφέρουμε στο Κανκούν, τότε ενδεχομένως τα καταφέρουμε σε κάποιο άλλο φόρουμ. Αυτό που εγώ θέλω να πω σε αυτούς είναι ότι αν δεν καταλήξουμε σε σημαντική πρόοδο στο Κανκούν, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για να καταλήξουμε σε κάποιο άλλο φόρουμ. Ποιο είναι το άλλο φόρουμ, το G20 θα είναι αυτό, το G8, το G2, Προσπάθησαν πέρυσι χωρίς αποτέλεσμα όμως. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλα τα συμβαλόμενα μέρη, όλες οι χώρες του G77 που ενδιαφέρονται για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή και που έχουν συμφέρον να καταλήξουμε σε πρόοδο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε αυτά αποτελέσματα στο Κανκούν. Διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα και με τα προγράμματα των ΗΕ. Εθνών και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτικό φόρουμ, θα ήταν πραγματικά καταστροφή να μην καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα στο Κανκούν. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να σημειώσουμε την απαραίτητη πρόοδο στο Κανκούν. Εγώ και οι ειδικέ μου υπηρεσίε θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε κυρία Επιτροπέ για τις εξηγήσεις αυτές πολύ πλούσιο σε περιεχόμενο αυτά που μας είπατε. Νομίζω ότι ε, σαφώς είναι προφανές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας υποσελίζει και στο ψήφισμά μας διευκρινίσαμε ότι ο ΙΕ θα πρέπει να είναι το πλαίσιο για διεθνείς συμφωνίες και όχι κάποιο άλλο πλαίσιο. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες διαπραγματευτικές οδοί, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκρίνησε ότι θα πρέπει να μείνουμε στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Και από εκεί βήμα προς βήμα να δούμε πώς θα γίνει και θα επιτευχθεί η πρόοδος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε στο Κανκούν. Αλλά ευχαρίστω σας προσκαλούμε και σε διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε την ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι το 4 υπαριθμών. Προφορική ερώτηση της Ελένα Οάννα Αντωνέσκου σχετικά με τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσω στη συνάδελφο το λόγο, αλλά λίγο, λίγο να περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα να ησυχάσει λίγο η αίθουσα. sich beruhigt haben oder vor die Tür gegangen sind. Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε. Σα uh, Σας παρακαλώ. Oh, Ξεκινήστε νομίζω, συνάδελφε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτά που... για όλα αυτά αυτό το θέμα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κρίμα που δεν έχουμε περισσότερους ε, συνάδελφους παρόντες, αλλά εντάξει, ίσως και στο μέλλον θα το εξετάσουμε και πάλι. Να σας παρουσιάσω ένα ιδιαίτερα αρνητικό πρόβλημα και έχει να κάνει με πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναφέρω την Ρουμανία, τη χώρα μου σαν ε, παράδειγμα. είχαν άνοιξα τα dream shops, τα καταστήματα πώληση ονείρων, δηλαδή νόμιμα, νόμιμες ναρκωτικές ουσίες ε, που είναι ε, υποκατάστατα βαρέων ναρκωτικών κοκαίνη, ροήνη, το έκσταση και που είναι απαγορευμένες για ανθρωπινή χρήση εδώ χρησιμοποιούνται, επαναλαμβάνω, για να προκαλέσουν ε, ε, τα ίδια που προκαλούν και οι παραπάνω επικίνδυνες ουσίες. Έχουμε 500.000 χρήστες ε, στη Ρουμανία. Το 5% του πληθυσμού είναι ανισχυτικός αυτός ο αριθμός και νέοι και κύριοι χρήστες ανάμεσα, έχουν ηλικίας ανάμεσα 14 και 23 και ε, δυστυχώς τώρα τελευταία είχαμε και πολλές περιπτώσεις θανάτων και ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται όλα ένα και περισσότερο. Spice ε, λέγονται έτσι γενικά αυτά τα προϊόντα και αυτές οι ψυχοτρόπες ουσίες ε, δημιουργούν ε, και διάφορα στους χρήστες που σε συνδυασμό και με παραγόγα ε, της Καναβέως. Εδώ τα μείγματα αυτά έχουν και, περιέχουν και βαρέα μέταλλα πολλές φορές και είναι προϊόντα που λένε ότι είναι φυσικά συμπληρώματα ε, και πολλές φορές πουλιούνται και σαν ε, αρωματικά άλατα <laughs> για το λουτρό, τι να σας πω τώρα. Εδώ δεν υπάρχει πολλές φορές έλεγχος στο πραγματικό περιεχόμενο αυτών των ουσιών. Μόνο βλέπουν και πιστεύουν αυτό που λέει η ετικέτα. Και πολλοί ψυχίατροι λένε ότι υπάρχει μια εξάρτηση που είναι υψηλότερη από της ηρωίνης και της κοκαίνης και ότι δημιουργείται αυτή η εξάρτηση από τις πρώτες φορές χρήσης αμέσως και οι αρχές της Ρουμανίας ε, μέσω ε, διατάγματος ακριβώς ε, κυβερνητικού πρότεινε η κυβέρνηση αυτές να είναι να θεωρούνται σαν απαγορευμένες εσπίσεις ουσίες. Και τον Απρίλιο ίσχυσε αυτός ο νέος νόμος, αλλά μετά από λίγο ε, άλλαξαν τα πράγματα και πάλι, τους ξέφυγε κατάσταση από τα χέρια και πολλές φορές εισάγονται προϊόντα και πολλές φορές έχουμε πολλούς συνδυασμούς παρομοίων ουσιών ε, που προκαλούν τα ίδια αποτελέσματα. Ψυχοτρόπες ουσίες λοιπόν ε, και η κατάσταση δυστυχώς έχει ξεφύγει επαναλαμβάνω από τα χέρια μας και η περίπτωση της Ρουμανίας ταυτόχρονα είναι ε, αρκετά ενδεικτική και ίσως άλλα κράτη δεν σημαίνει το ίδιο. Τέλο πάντων αυτά τα νέα προϊόντα είναι νέος κατάλογος ουσιών και είναι αδύνατο να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα οι αρχές γιατί μέχρι να κυκλοφορήσουν αυτές τις καινούριες ουσίες, αυτά τα καινούργια παράγωγα και να μπουν στην απαγορευμένη ε, στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών περνάει καιρός και κινδυνεύει κόσμος. Εδώ λοιπόν ε, θα πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε το φαινόμενο. Δύσκολο είναι πάντως αυτός ο τρόπος με το συμπερίληψη δηλαδή στον κατάλογο ε, απαγορευμένων σιών. Εδώ το θέμα δεν νομίζω ότι είναι μόνο της Ρουμανίας αλλά της Ευρώπης γενικά. Χρειάζεται να λάβουμε πρωτοβουλίες. Γι' αυτό το λόγο ζήτησα από την Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα και να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, η πώλησή τους, ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει σχετικά η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφα Αντωνέσκου. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Αυτό το οποίο πλήττει πολλές χώρες, χώρες και κυρίως πάρα πολλούς νέους να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Έχουμε δύο δυνατότητες, δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ε, Γενική Διεύθυνση, από την Υπηρεσία για τα Ναρκωτικά και δεν ξέρω ποιος θα πάρει πρώτο το λόγο. Thank you, Chairman, for giving me the floor. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση δικαιοσύνης και με μόνη μου γιατί ο συνάδελφος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και να ευχαριστήσω την κυρία Αντωνέσκου που έθεσε το ερώτημα αυτό το οποίο είναι πραγματικά πολύ εύστοχο για μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην... σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά. Η κατάργηση των ναρκωτικών αποτέλεσε το βασικό θέμα τα τελευταία χρόνια, τα legal highs όπως τα λένε. Πρόκειται για, βοτανι... για βότανα συνθετικά ναρκωτικά τα οποία χρησιμοποιούνται όλο και παραπάνω, όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πάρτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθούνται ως άλατα για το λουτρό, ως... Ε... για τα φυτά, σας δίνω κάποια παραδείγματα, αλλά προφανώς ε, και σαφέστατα προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Ιδιαίτερα δημοφιλή επειδή ε, εμπορεύονται ως νόμιμα. Είναι μια νόμιμη εκδοχή σε διάφορων άδων παράνομων ουσιών και ο κόσμος θεωρεί ότι εφόσον είναι νόμιμα είναι και ασφαλή. ή εν θεωρεί ότι δεν είναι παράνομος ο χρήστης. Είναι ο νόμος νόμιμα. Δεν απαγορεύονται. Δεν απαγορεύονται επειδή είναι καινούργια και τα γνωρίζουν ακόμα οι αρχές τα κρατη σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο. Αλλά οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, ο κίνδυνος που παρουσιάζουν στην υγεία, είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος. Πώ το αντιμετωπίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχά, μπορεί να υπάρξει απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο των ουσιών αυτών. Τα κράτη-μέλη επίση είναι αρμόδια για την νομοθεσία, για τη λειτουργία των shops αυτών, των drink shops, των καταστημάτων που πολλούν τα νέα αυτά ναρκωτικά. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να υπάρξει αποτελεσματικότητα σε εθνικό επίπεδο αν οι πολίτες μπορούν να βρουν το ίδιο ναρκωτικό είτε στο ίντερνετ είτε σε μια διπλανή χώρα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των νέων ναρκωτικών. Μιλάμε για την απόφαση 387 του 2005 που επιτρέπει και οργανώνει την αλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις νέε ψυχοτρόπε αυτές ουσίε. Βάσει τη απόφαση του Συμβουλίου αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση σύντομα για το πώ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η μεθατρόνη, μια ολοένα και πιο δημοφιλή ουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προ το παρόν απαγορεύεται στα 14 κράτη-μέλη. Η έκθεση αξιολόγηση κινδύνου της Υπηρεσίας ε, για τα Ναρκωτικά στη Λισαβόνη καταδεικνύει ότι η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολογούν την εφαρμογή της απόφασης αυτής του Συμβουλίου για τα νέα ναρκωτικά αυτά. Ξεκίνησε η αξιολόγηση πριν το καλοκαίρι και θέλουμε να την ολοκληρώσουμε μέχρι τα μέσα του 2011. Βάσει των πορισμάτων της ε, αξιολόγησης αυτής θα υποβάλουμε νομοθετικές προτάσεις για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του οργάνου αυτού, για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το ταχαίο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και την ταχαία μεταβαλλόμενη αγορά των ναρκωτικών. Τι εξετάζουμε λοιπόν. Θα εξετάσουμε τη νομική βάση καταρχάς της απόφασης του Συμβουλίου. Είναι ε, εργαλείο του τρίτου πυλώνα και θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και φυσικά θα πρέπει να δοθεί ρόλος και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται βάσει του εργαλείου αυτού προς το παρόν. Το, συμβούλιο, το Κοινοβούλιο βάσει της νομοθεσίας του 2005 δεν έχει τέτοια δικαιώματα. Κατά δεύτερον θα κοιτάξουμε τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί τέσσερις φάσεις από ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών μέχρι κοινή έκθεση για ένα νέο ναρκωτικό από την υπηρεσία στη Λισαβόνια και στην τη Europol. Τρίτον, έκθεση αξιολόγησης κινδύνου από την υπηρεσία στη Λισαβόνα και τέλος ε, η τελική πολιτική. Θα κοιτάξουμε πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν ε, τα στάδια αυτά και πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι ανάλογες προθεσμίες. Και επίσης θα εξετάσουμε κατά πόσον ο νομικός τρόπος αντιμετώπισης των νόμιμων ψυχοτρόπων είναι σωστός. Επειδή είναι τόσο γρήγορα μεταβαλλόμενη η αγορά, μπορέσουμε να, θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε ίσως ομάδες ουσιών. Ίσως να υπάρχουν διάφορες ε, δυνατότητες ελέγχου. Γιατί προς το παρόν δεν έχουμε ενδιάμεσες λύσεις, για παράδειγμα. Επίσης, να σας πω ότι οποιαδήποτε νέο εργαλείο θα ακολουθήσει τις ε, αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Άρα, οποιαδήποτε εργαλείο θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και θα πρέπει να είναι ισορροπημένο, λαμβάνοντας υπόψη πτυχές όπως και η δημόσια υγεία, αλλά και ο σεβασμός των διεθνών συμβάσεων. Εξετάζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας και φυσικά θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε σε οποιαδήποτε φάση θεωρήσετε ότι χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος, για τις απαντήσεις. Η συνάδελφος Αντωνέσκου ε, έχει να κάνει και άλλα ερωτήματα. Uh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία για όσα μας είπε για το θέμα αυτό και χαίρομαι που ακούω ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ε, την ε, εφαρμογή της οδηγίας 2005 την 388 ε, για τις εκτιμήσεις ε, για αυτές τις ουσίες ε, και ότι θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο μιας ε, συνεχούς παρατήρησης και για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη μας κατά του φαινομένου αυτού θα πρέπει να αλλάξει η μέχρι τώρα στάση μας. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε νέα μέτρα, να έχουμε νέες ρυθμίσεις αυτά τα spices, αυτές οι νέες ουσίες ε, βλέπουμε ότι συνεχώς βγαίνουν και κυκλοφορούν στην αγορά με καινούρια μορφή, με καινούριες ε, συνθέσεις ε, συνθετικά προέρχονται από την κάναβη που αποτελεί τη βάση πολλές φορές ε, και γι' αυτό ακριβώς είναι πάντα επικίνδυνες και χρειάζονται μια εκτίμηση κινδύνου. Αυτό που αναρωτιόμαστε εμείς τώρα η σημερινή ρύθμιση, κατά πόσο είναι αποτελεσματική έτσι επιτόπου, αν λάβουμε υπόψη μας το φαινόμενο αυτό, γιατί βλέπουμε αυτές τις ε, ε, τα προϊόντα σύνθεσης, αυτές τις χημικές ουσίες ε, και μέσω του ίντερνετ ότι εμφανίζονται σαν νόμιμες. Τι, έγινε, τι γίνεται, ταυτόχρονα αποδεικνύουν ότι αυτή η αγορά έχει τεράστιες δυνατότητες για καινοτομίες και δημιουργία νέα προϊόντα. Και ε, αυτό σημαίνει ότι αποτελούν για μας ιδιαίτερη επίσης πρόκληση. Θα πρέπει να εξετάσουμε κάθε μία ξεχωριστά ουσία από αυτές, αλλά το τι προσθέτουμε σιγά σιγά στον κατάλογο των απογραφημένων δεν αποτελεί κατά την απόψή μου λύση. Είναι πολύ άριθμες αυτές οι ουσίες προϊόντα σύνθεσης. Δεν έχουν ρυθμιστεί μέχρι τώρα οι πωλήσει τους και αποτελούν κίνδυνο, επαναλαμβάνω. Θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και χρειάζεται μελέτη του προβλήματος και ελπίζω να μας υποστηρίξει η Επιτροπή Περιβάλλοντος επίσης για την λήψη μέτρων. Είναι δεινό το πρόβλημα και βλέπουμε το όλα και περισσότερο διονγκώνεται αυτό το πρόβλημα στις διάφορες χώρες μας και γι' αυτό θα πρέπει ακόμα πιο ιδιαίτερα να μας ανησυχεί. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε την συνάδελφο Έχουμε την έκθεση για τη Ρουμανία και τις ουσίες αυτές. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ε, χώρες. Είναι διεθνής η αγορά σε ό,τι αφορά την εμπορία και την κατασκευή, την παρασκευή των ε, ουσιών αυτών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονισμένα να δράσει με συγκεκριμένες ε, κατευθυντήρες γραμμές. Σας ευχαριστώ λοιπόν που θέσατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε σχετικές δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν θεωρεί ότι καλύφθηκε. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε και το λόγο. Να απαντήσω και στην ερώτηση αυτή. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας για την καταπολέμηση αυτών των νέων ναρκωτικών είναι όντως το ζήτημα αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει. Η κυρία Αντωνέσκου αναφέρθηκε στο ότι αυτή τη στιγμή απαγορεύουμε τις ουσίε μάλλον ουσίες μία προς μία, το οποίο ενδεχομένως να είναι αναποτελεσματικό και να καταναλώνει πάρα πολύ χρόνο. Άμα σκεφτεί κανείς ότι μία ουσία που χρησιμοποιείται σήμερα θα αντικατασταθεί από μία παρόμοια ουσία στο μέλλον, κάνοντα απλώ μια μικρή αλλαγή στην σύσταση τη ουσία αυτή. Επομένω, θέλουμε να δούμε αν γίνεται από νομική πλευρά να απαγορεύουμε πλέον ολόκληρε ομάδε ουσιών και όχι ξεχωριστέ ουσίε πλέον. Αυτό είναι ένα μόνο από τα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Οι προθεσμίες επίσης είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα. 14 κράτη-μέλη έχουν απαγορεύσει τη μεθοδρόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την επόμενη εβδομάδα την πρότασή της για το πώς να αντιμετωπιστεί η ουσία αυτή. Από την άλλη, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τα επιστημονικά δεδομένα προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια πολιτική απόφαση. Καταλαβαίνετε ότι ε, καλούμεθα εμείς να δώσουμε απάντηση σε κάποιες πολύ πολύπλοκες ε, ερωτήσεις. Πάντως το νέο αυτό μέσο που θα έχουμε θα το παρουσιάσουμε στις αρχές του επόμενου έτους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Uh, uh, να κλείσουμε λοιπόν και το σημείο αυτό και να περάσουμε στο επόμενο, το οποίο είναι το 5 της ημερήσιας διάταξης, Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντικο-Οικονομική Λογαριασμή. Ε, μια έκθεση που ξέμεινε στα δικά μου χέρια, που όμως με ενδιαφέρε ιδιαίτερα και χάρηκα που την κατήρτισα, γιατί το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς ε, διαμορφώνεται η περιβαλλοντική πολιτική στα κράτη-μέλη της Ένωσης, κατά πόσον σημειώνονται επιτυχίες ή όχι. Έχουμε όλες τις συλλογή στοιχείων για τις οικονομικές δραστηριότητες, αλλά δεν έχουμε σχετικά στοιχεία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν καλώς ορίζει το γεγονός ότι ανέλαβε την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση. Για τις περιβαλλοντικούς εθνικούς λογαριασμούς, όπως αναφέρονται στην έκθεση. Υπάρχει συλλογή στοιχείων σε κάποιους τομείς και τα κράτη-μέλη σε θελούσια βάση μπορούν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία τέτοια μέσω της ε, Ευρωστάτ και κατά την ε, οικονομική κρίση σημειώθηκε μία τάση αναστολής ή περιορισμού της διαδικασίας αυτής. Άρα νομίζω ότι σωστά απάντησε έτσι η περιορισμου τη διαδικασια αυτη αρα Επιτροπή προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η παροχή των στοιχείων αυτών. Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε τρεις ενότητες της ε, λογαριασμού για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους φόρους για το περιβάλλον και το συνολικό υλικό. Τρεις τομείς λοιπόν. Άκουσα συζητήσεις από σχετικές υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με τέτοια θέματα σε εθνικό επίπεδο και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες ενότητες. Είναι σωστό ίσως αρχικά να ξεκινήσουμε από την κατεύθυνση αυτή, αλλά θα ήθελα να προσθεθούν και άλλες ενότητες όπως το νερό, οι περιβαλλοντικές επιδοτήσεις και άλλες ενότητες. Όλα αυτά θα πρέπει να προσθεθούν προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η εικόνα που θα λαμβάνουμε. Επίσης, θα πρέπει να εμπεριλαμβάνονται μόνο τα χρησιμοποιημένα υλικά, αλλά και τα μη χρησιμοποιημένα υλικά. Μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο υλικών που δεν χρησιμοποιούνται. Απορρίψεις, για παράδειγμα, στην αλία, στις εξορίξεις. Μη χρησιμοποιηθέντα μη μεταλλικά υλικά. Αυτά τα στοιχεία δεν χορηγούνται και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβανόντουσαν σε, μια τέτοια, σε ένα τέτοιο συνολικό λογαριασμό. Άνοιξα λοιπόν την πόρτα προκειμένου σε εθελοντική βάση να συμπεριληφθούν οι ενότητες αυτές. Γιατί ίσως αυτό να συνεπάγεται για κάποιες χώρες σε ένα μεγάλο φόρτο σημαντικό είναι αν θέλουμε να υπάρχει ένας τέτοιος περιβαλλοντικός λογαριασμός να το γνωρίζουν αυτό οι διάφοροι παράγοντες αλλά και οι πολίτες. Ξέρουμε ότι υπάρχει το ετήσιο ΑΕΠ. Πρόκειται για μία παράμετρο η οποία, η οποία χρησιμοποιείται σε πολιτικές συζητήσεις αλλά δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με το λογαριασμό αυτό τον περιβαλλοντικό, κατά πόσο είναι θετικός ή αρνητικός. Ίσως και αυτός θα έπρεπε να δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Και επειδή τα πράγματα αυτά εξελίσσονται διαρκώς, θετικό η Ευρωπαϊκή αυτό θα επρεπε να κάνει μια αναθεώρηση των στοιχείων που συλλέγονται. Να γίνεται δηλαδή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε τρία χρόνια με ενδεχόμενες τροποποιήσεις και προσαρμογές για να βελτιώνεται το εργαλείο αυτό. Αυτό εν συντομία ήταν το περιεχόμενο της έκθεσης της οποίας ε, κατήρτισα. Έχουμε μαζί μας και τους σκιώδεις εισηγητές. Merci, Monsieur Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν έχω και πολλά να πω. Ε, είναι πραγματικά αξιόλογη εργασία σα Καμία τροπολογία, εκτό αν ε, κάνουμε κάτι όταν την ε, διαβάσουμε και πάλι. Πάντω θα ήθελα να συγχαρώ για αυτή την εργασία και συμφωνώ με αυτέ τι τροπολογίε που προτείνετε ενδεχόμενα. Είναι λογικέ σαν τροπολογίες, αλλά λοιπόν προ στιγμή δεν μπορώ να σα προσάψω τίποτα, ούτε να αλλάξω κάτι και αυτά και σα ευχαριστώ. Μάλιστα, πολύ καλό αυτό. Πάντα χαίρεται ένα εισηγητή να ακούει τέτοια σχόλια. Ο κύριο Σνέλχαρτ, ναι, δεν είμαι σκιώδη. Δεν ξέρω ποιο είναι σκιώδη από την ομάδα μου, αλλά θεωρώ ότι μάλλον είναι κάπως επικριτική η στάση μου για το θέμα αυτό, γιατί οι προτάσει του Προέδρου βασίζονται στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημειώνω αυτό. Και επίση θεωρώ ότι κοιτώντα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σωστό είναι. Σωστές είναι οι τροπολογίε που υπέβαλε ο Πρόεδρος. Αναρωτιέμαι όμως, τι θα, μας, ε, τι θα κερδίσουμε αν με τόση γραφειοκρατία συλλέξουμε πληροφορίες προς αξιολόγηση. Ποια θα είναι τα πορίσματα που θα εξαγάγουμε από τις πληροφορίες αυτές. Εγώ αυτό που ζητάω πάντα είναι το εξή. Θέλουμε να υπάρχουν, θέλω να υπάρχουν λίγες παράμετροι οι οποίοι θα καλύπτουν όμως πολλά. Έχουμε την νομοθεσία για την ατμόσφαιρα και την του της ατμόσφαιρας για τα ύδατα. Υπάρχει δεσμευτική νομοθεσία στα κράτη-μέλη την οποία και εφαρμόζουν. Σε καμία άλλη περιοχή του κόσμου δεν υπάρχει τόσο νομοθεσία για το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα τα κάνει τα στοιχεία αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και άλλους λογαριασμούς. Με αρνητική αξιολόγηση. Τι θα γινόταν αν δεν είχαμε υπερβολικά αυστηρούς κανόνες. Πώς θα όταν τότε η κατάσταση. Να το κοιτάξουμε και αυτό. Ή ποια θα πρέπει να είναι η απόδοση της βιομηχανίας για να εφαρμόσει αυτά τα οποία αποφασίζουμε εδώ. Όλα αυτά τα ερωτήματα πάντα ανακύπτουν στο δημόσιο διάλογο και πάντα βασανίζουν το ευρύ κοινό, γιατί ακριβώς αυτά είναι τα σημαντικά για τον κόσμο. Γιατί αν συλλέγουμε στοιχεία και λέμε «Α, τι άσχημα που πάνε τα πράγματα», θα πρέπει να εφαρμόσουμε πιο αύστηρη νομοθεσία τι θα κερδίσουμε. Αν συλλέγουμε όμως τα στοιχεία για να υπάρχει μια συγκρισιμότητα μεταξύ των κρατών μελών, για να δούμε ποια κράτη-μέλη δεν εκπλήρωσαν τις ε, αυστηρές προδιαγραφές, τότε μάλιστα, τότε θα καταλάβαινα ότι συλλέγουμε τα στοιχεία αυτά, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί πολλά κράτη μπορεί να θεωρούν ότι ε, δεν πάνε να σας ζητάνε οι άλλοι, εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε. Άρα, να σας ε, προειδοποιήσω και να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Να μην ξεκινήσουμε να κάνουμε την νομοθεσία όλο και πιο αυστηρή. Ευχαριστώ, συνάδελφε Σνέλχαρτ. Θα πω δύο λόγια, μετά ο Κρήτονας θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η τροπολογία 8 που ζητά τη δημιουργία περισσότερων κατηγοριών στον κανονισμό και αναφέρεστε συγκεκριμένα στο νερό καθώς επίσης και στους δασοκομικούς λογαριασμού. Γίνεται επίσης αναφορά στην ξυλία θα ήθελα να προσθέσουμε δύο ακόμα σημεία στο παράρτημα 3. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν αρκετές διατάξεις για τη συλλογή δεδομένων για το νερό. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να προβλέπετε στο παράρτημα 3, γιατί αναφερόμαστε εδώ πέρα στα δεδομένα τα οποία πρέπει να υποβάλλονται στα πλαίσια τις οδηγίες πλαίσιο για το νερό. Επίσης, τα αλληλευτικά αποθέματα θα πρέπει επίσης να αναφέρονται, ενδεχομένως στο παράρτημα 3. Στο παράρτημα 1 τώρα, όπου αναφερόμαστε στους λογαριασμούς για την ατμόσφαιρα, αναφέρεστε εδώ πέρα στο UNCCC, αλλά δεν δημιουργείται υποκατηγορίες όσον αφορά τις πηγές εκπομπών, όπως προβλέπεται από την σύμβαση αυτή. Επίσης, μολονότι τα κράτη-μέλη ήδη υποβάλλουν δεδομένα στα πλαίσια του LULUCF, αλλαγή στη χρήση της γης και χρήση της γης, δεν περιλαμβάνουν τα δεδομένα αυτά, ενώ θα μπορούσαν να προβλέπονται στο παράρτημα 1. Γιατί αργότερα θα αναγκαστούμε να συμπεριλάβουμε αυτά τα δεδομένα. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε τώρα λοιπόν από την αρχή. Ähm, Ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μας πει γιατί συλλέγουμε τα στοιχεία αυτά. Ποιος είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Είναι μήπως από την Ευρωστάτ είναι κάποιος. Thank you very much for giving the opportunity to uh, uh, σας ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσετε την πρόταση αυτή στην, Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή σας. Να απαντήσω καταρχάς σε κάποια σχόλια και τις ερωτήσεις. Και μετά θα περάσω σε κάποιες από τις τροπολογίες. Καταρχάς, να σας δώσω το υπόβαθρο και το ιστορικό της πρότασης αυτής. στην Ευρωστάτ. Εργαζόμαστε και δουλεύουμε για τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς εδώ και χρόνια. Κάναμε πληροτικές μελέτες και αναπτύξαμε μία μέθοδο που είναι απαραίτητη για να μπορέσουν οι χώρες να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά βάσει μιας στρατηγικής την οποία ενέκριναν οι γενικοί διευθυντές το 2008. Η στρατηγική αυτή περιελάμβανε διάφορα βήματα για την εφαρμογή των λογαριασμών. Και οι τρεις ενότητες οι οποίες ε, επικράτησαν είναι αυτές που σας παρουσιάζουμε εδώ σήμερα. Αυτά τα στοιχεία συλλέγονται ήδη σε θελούσια βάση. Και έτσι η δυσκολία συζήτησης ε, με διάφορες χώρες και της υποστήριξης ε, εκ μέρους των χωρών δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν γίνεται σήμερα συζήτηση στο Συμβούλιο η οποία όμως εξελίσσεται ομαλά και αναμένουμε ότι δεν πρόκειται να προκύψουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά εν είδη εισαγωγής. Για να μιλήσουμε τώρα για τη σημασία των περιβαλλοντικών λογαριασμών και τις δυνατότητες που συνεπάγονται για την οικονομική ανάλυση του περιβάλλοντος και τη σχέση που υπάρχει με την οικονομία, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σύστημα οικονομικών εθνικών λογαριασμών, το οποίο ισχύει εδώ και χρόνια, και οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί είναι η σύνδεση με τους ε, οικονομικούς λογαριασμούς. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό και το εργαλείο αυτό για την οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση, γιατί επιτρέπει, για παράδειγμα, να εξετάσουμε τα διάφορα αποτελέσματα για τις εκπομπές της ατμοσφαιρικές, για παράδειγμα, και να υπάρξει και σύνδεση με τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Άρα συνδέεται η εκπομπή όχι με την παραγωγή μόνο, αλλά και με την κατανάλωση. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι η σχέση μεταξύ της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των εκπομπών. Υπάρχει δυνατότητα τέτοιας ανάλυσης μέσω των περιβαλλοντικών λογαριασμών. Αυτή είναι η ισχύ ε, του συστήματος και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει σχετική νομοθεσία, γιατί υπάρχει δυνατότητα σύνδεση των στοιχείων αυτών κατά ένα αρμονισμένο τρόπο. Και της ε, δίνεται δυνατότητα ανάλυσης σημαντικής για τις ε, περιφερειακές μελέτες. Έτσι λοιπόν δικαιολογείται το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το σύστημα αυτό. Και όπως είπα, ο λόγος που κινούμαστε βαθμιδών σταδιακά είναι ακριβώς επειδή το κόστος είναι υψηλός, υψηλό και είναι διαφορετικό το επίπεδο των διαφόρων κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε έτσι βαθμιαία. Αυτά ήθελα να διευκρινίσω. Να αναφέρω επίσης δύο συγκεκριμένες τροπολογίες τις οποίες προτείνει ο εισηγητής οι 8 και οι 9. για την 8, όπως είπα, συμφωνούμε απόλυτα ότι τα τρία αυτά στοιχεία τα οποία παρουσιάζουμε σήμερα στο σχέδιο της πρότασης αποτελούν ένα τμήμα μόνο μια συνολικής στρατηγικής που αποδέχτηκαν το 2008 οι γενικοί διευθυντές. Υπάρχει μεν η συμφωνία, αλλά θεωρούμε ότι το να συμπεριληφθούν αυτά στο κείμενο όπως προτείνεται στην τροπολογία 8 θα είναι δύσκολο και δεν θα το αποδεχτούν οι χώρες. Μπορούμε να το σημειώσουμε αυτό ότι υπάρχει αυτή η στρατηγική και να το συμπεριλάβουμε ως εκτιμώντας στην αρχή του κειμένου. Να πούμε δηλαδή ότι έχουν συμφωνήσει οι γενικοί διευθυντέ του NSI να υπάρξει μια βαθμιαία προσέγγιση. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να πω για τις τροπολογίες. Για την τροπολογία 9 τώρα. Όπως σας είπα εξ αρχής, κάνουμε κάποιες πιλωτικές μελέτες και τώρα έχουμε ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα πιλωτικών μελετών για να κινηθούμε παραπάνω, περαιτέρω στον τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και προϊόντων. Το να συμπεριληφθεί όμως κάτι εδώ, ίσως να είναι αντιπαραγωγικό και ίσως να προκαλέσει αντίδραση κρατών μελών. Θεωρούμε λοιπόν ότι ίσως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε ένα εκτιμώντας πάλι το ποια είναι η πρόθεσή μας για το μέλλον. Ίσως αυτό να επαρκεί και να καταστήσει το κείμενο πιο αποδεκτό από τα κρατημέλη. Για να κλείσω, θεωρούμε ότι είναι σύντομο να εφαρμοστεί σύντομα η νομοθεσία αυτή, γιατί τις χρειαζόμαστε ήδη τις πληροφορίες αυτές και είναι σημαντικό να υπάρχει νομική βάση. Όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και λυπάμαι που δεν είπα καλά το όνομά σας Σας ευχαριστούμε και για την εργασία που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια σε εθελοντική βάση ο συνάδελφος με ρώτησε, ο συνάδελφος Σνέλχαρτ ρώτησε κάτι. Θα ήθελα να σας πω ότι με, την, με τα στοιχεία αυτά δεν θέλουμε απλά να μειώσουμε και να πούμε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των κρατών μελών. Όχι. Θέλουμε να διαπιστώσουμε αν έχει επιτυχία η περιβαλλοντική μας ε, πολιτική ή αν θεωρούμε μόνο ότι είναι επιτυχής η πολιτική ως προς το περιβάλλον. Μακροπρόθεσμα θέλουμε να βελτιωθούν τα πράγματα, όχι να επιδεινωθούν. Και δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να το κρίνουμε αυτό. Για τις ερωτήσεις του κυρίου Αρσένη. Να τις κοιτάξω, αλλά ακούω ότι τα στοιχεία για το νερό και για τις εκπομπές συμπεριλαμβάνονται ήδη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στο 3α επίσης το καινούριο ζητούνται τα στοιχεία αυτά. Αλλά θέλει κάτι να ρωτήσει ο συνάδελφος Σνέλχαρτ. Ναι, αυτό που με ανησυχεί στην όλη ιστορία είναι το εξή. Θέλουμε πάλι να συλλέξουμε στοιχεία και υποθέτω ότι κινούμαστε προς την κατεύθυνση του 2014 και 2019 να δημιουργηθούν νέες παράμετροι για τις επιδοτήσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί ποτέ σε τόσο, χρονικό, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε, να συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Λέμε για παράδειγμα, κάποιοι λένε ότι θέλουμε 10 χρόνια για να αποσβεστεί μια αιωλική τουρμπίνα. Είναι πραγματικά συσήφιο το έργο για να συλλεχθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές. Μπορούμε να καταρτήσουμε τέτοιες λογαριασμούς, αλλά ειλικρινά θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Δεν ξέρω, μπορεί να με πείσει ο εισηγητή στην πορεία. Ναι, θα το επιχειρήσω, συνάδελφε. Δεν έχετε αντιρρήσεις κι εσείς να συλλέγονται οικονομικά στοιχεία από όλες τις επιχειρήσεις που καταγράφουν με ακρίβεια τους κύκλους εργασιών, τις εξαγωγές, τις εισαγωγές, όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία τα γνωρίζουμε. Τα οικολογικά στοιχεία εν μέρη δεν τα γνωρίζουμε. Και σκοπός, επαναλαμβάνω, είναι απλά να δημιουργηθεί μια βάση για το κατά πόσον σημειώσαμε επιτυχία ή αποτυχία με την πολιτική που ακολουθήσαμε. Για αυτά που μας είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωστάτου. Εντάξει, στο 8, στην τροπολογία 8 προτείνω επιπλέον ενότητες. Αναφέρω όμως αναπτύσσει ως προτεραιότητα τα εξή στοιχεία. Δεν αναφέρω το 2013 ή το 2014. Στην τροπολογία 11 αναφέρουμε ότι μετά από 5 έτη η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει έκθεση εφαρμογής και να υποβάλει ενδεχόμενες βελτιώσεις. Πρόκειται για ένα νομοθετικό πλαίσιο δεν σημαίνει αυτό ότι όλα θα λειτουργήσουν 100%. Μετά θα το ακούσουμε αυτό, φαντάζομαι, στην ε, έκθεση εφαρμογής. Μάλιστα. Uh, Παίρνω και πάλι το λόγο κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η έκθεση είναι πολύ καλή και θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι ε, αναφέρονται όντως εκπομπές στο παράρτημα 1, αλλά αυτό το οποίο ζητάω εγώ είναι να υπάρχουν ε, διατάξεις για υποκατηγορίες όπως έχουμε να έχουμε υποκατηγορίες στις α, εκπομπές, όπως προβλέπονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, το ίδιο και για το Ίδωρ, Στο άρθρο 3α, το νέο, λέγεται ότι πρέπει και άλλες μέθοδοι να αναπτυχθούν. Αυτό που λέω ουσιαστικά είναι ότι θα πρέπει να έχουμε διατάξεις για τη συλλογή δεδομένων ειδικά για το νερό, πέρα από τους γενικούς μηχανισμούς προβλέπονται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ενδεχομένως δηλαδή να επισέλθουμε εμεί σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως τα περισσότερα στοιχεία βρίσκονται ήδη και η έκθεσή σας είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ. Για τα στοιχεία για το νερό. Υπάρχει κάτι από την σχετική οδηγία. Τι κάνουμε με το νερό. Yeah, uh, Όσον αφορά το νερό, Έχουμε τις πληροφορίες συλλογής από την οδηγία πλαίσιο, συλλέγονται οι πληροφορίες αυτές. Τώρα όμως τις ενότητες που θέλουμε να πτύξουμε στο μέλλον θα υπάρχει και μία ενότητα ξεχωριστή που θα φέρει το όνομα Λογαριασμή ύδατος και θα μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για την οικονομία του νερού. Πολύ πιο πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά το νερό που δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή. Όπως σας είπα όμως ε, η οδηγία πλαίσιο για το νερό προβλέπει ήδη μια κάποια συλλογή πληροφοριών για το νερό που συλλέγονται αυτή τη στιγμή από τη Eurostat ή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. And it's exactly data that we want to be put... Και ακριβώς αυτά τα δεδομένα θέλουμε εμείς στο παράρτημα. Τα έχουμε τα δεδομένα αλλά συμπεριληφθούν στο παράρτημα. the, uh, sorry, the question is Το αν θα συμπεριληφθούν τα στοιχεία αυτά στο MFA θα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα φορτίσει πάρα πολύ το όλο σύστημα και δεν θα καταφέρει το σύστημα να λειτουργήσει σωστά. Δεν θα είναι δυνατό, τουλάχιστον στη φάση αυτή, να συμπεριληφθούν τα στοιχεία αυτά. Οι συνάδελφοί μου πάντως μου λένε ότι θα έχουμε σίγουρα λογαριασμούς ύδατος. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δοκιμάσουμε το σύστημα αυτό για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του νερού με τον πιο περιεκτικό τρόπο. Η κυρία Παντολεύσκα είναι υπεύθυνη για τέτοια θέματα, για τους λογαριασμούς για το νερό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από μεθοδολογικής άποψης το είδωρο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν το συγκρίνουμε με την άλλη ροή υλικών που έχουμε μέσα στην οικονομία, το νερό έρχεται πρώτο. Αν δείτε λοιπόν τα δεδομένα, ένα μεγάλο τμήμα θα απασχολεί το νερό και όλα τα υπόλοιπα, μεταλλικά στοιχεία, μέταλλα κτλ. θα αντιστοιχούν σε ένα πολύ μικρό τμήμα τελικά του παραρτήματος με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε μια καλή συγκριτική αξιολόγηση όλων αυτών των υλικών που ρέουν μέσα στην οικονομία. Η Eurostat λοιπόν πιστεύει ότι για το νερό θα πρέπει να προβλέπονται ξεχωριστοί λογαριασμοί ύδατος. Δεν θα πρέπει το νερό δηλαδή να περιλαμβάνεται στους λογαριασμού για τη ροή υλικών. Και ακριβώς επειδή συμφωνούμε μαζί σας ότι το νερό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να μείνει εκτός. Και γι' αυτό σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στην ε, απαραίτητη μεθοδολογική οριμότητα που θα μας επέτρεπε να συμπεριλάβουμε το νερό στις ενότητες που προβλέπονται. Θα χρησιμοποιήσουμε πάντως τα δεδομένα τα οποία ήδη προβλέπονται και συλλέγονται στην οδηγία πλαίσιο για το νερό. Αυτά έχω να πω για το νερό. Να απαντήσω και την ερώτησή σας για τις εκπομπές. Η όλη λογική των περιβαλλοντικών λογαριασμών είναι να έχουμε μία κατηγοριοποίηση βάσει οικονομικής δραστηριότητας. Επομένως δεν γίνεται διαφοροποίηση των εκπομπών με βάση την πηγή τους, όπως κάνουμε για παράδειγμα σε διάφορους άλλους καταλόγους. Αυτή είναι η βασική διαφορά, αν θέλετε, ανάμεσα στους υφιστάμενους καταλόγους και τους καταλόγους που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μία κατηγοριοποίηση, όπως σας είπα, όχι με βάση την πηγή, αλλά με βάση την οικονομική δραστηριότητα. Αν πάρουμε τις μεταφορές, μεταφορές έχουμε στη γεωργία, στην εξωτερική βιομηχανία, στη μεταποίηση. Επομένως, τους καταλόγους έχουμε απλώς τον τίτλο «Μεταφορές» και βρίσκουμε όλες αυτές τις μεταφορές σε αυτόν τον κατάλογο. Στους δικούς μας λογαριασμούς, όλα αυτά τα δεδομένα θα είναι διαφοροποιημένα με βάση την οικονομική δραστηριότητα. Δεν θα γίνεται δηλαδή διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση με βάση την πηγή. Η όλη λογική που διέπει την προσπάθεια αυτή είναι τελώς διαφορετική. Σας ευχαριστώ. Θα κάνεις άλλο το λόγο. Ο κύριος Φλόρενς, ναι. Ήθελα να εκφραστώ και να εκφράσω την ε, υποστήριξή μου προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συλλογή στοιχείων, αλλά τι χρησιμεύουν όλα αυτά αν τα κράτη-μέλη δεν τηρούν τις δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι διάφορες οδηγίες. Υπάρχουν τρία-τέσσερα κράτη-μέλη από τα παλιά κράτη-μέλη, τα εντρετικά κράτη-μέλη, τα οποία δεν διαθέτουν μόνιμα τα στοιχεία αυτά, ούτε εφαρμόζουν την νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα κατά εξαίρεση να υποστηρίξω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ σήμερα και να πω το εξή θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερο δικαίωμα πρόσβαση στα δεδομένα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου εμείς να μπορούμε να καταρτίζουμε τα στατιστικά στοιχεία και να μπορούμε να κρίνουμε αν λειτουργεί ή όχι μία νομοθεσία. Θεωρώ ότι αυτή η νομοθεσία των τριών E, του triple E, δεν λειτουργεί επειδή δεν υπάρχουν ε, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Ε, πώς να παραπονιόμαστε λοιπόν και να ζητάμε παραπάνω. Αν θέλουμε λοιπόν τέτοια στοιχεία, να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποιο εργαλείο μπορεί να πάρει τα στοιχεία που χρειάζεται. Γιατί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα απόβλητα είναι μεγάλη η αποτυχία. Αυτό που κάναμε ήταν μια καλή νομοθεσία και τελικά δεν θέλω να κατανομάσω τι γίνεται. Να κάνουμε πιο λίγα, αλλά ό,τι κάνουμε να το κάνουμε καλύτερα. Και τι γίνεται με την παροχή τέτοιων δεδομένων σε ό,τι αφορά τα παλαιά ή τα καινούργια κρατημέλη. Ρωτάει ο Πρόεδρος, λαμβάνετε τα στοιχεία αυτά που θέλετε ή είναι αποσπασματικά τα πράγματα. there Κοιτάξτε, οποτεδήποτε υπάρχει μια νομική πράξη, οποτεδήποτε καταρτίζεται μια νομική πράξη για την συλλογή στατιστικών δεδομένων, τότε συνήθως λαμβάνουμε τα απαιτούμενα αυτά δεδομένα. Πάντα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν παρέκκληση και ενδεχομένως ότι χρειάζονται την περίοδο αυτή για να προετοιμάσουν και τα συστήματά τους. Στο τέλος πάντως περίοδου αυτής πάντα συλλέγουμε τα δεδομένα. Κάνουμε επίσης μία εποπτεία παρακολούθηση εφαρμογής των ε, νομοθεσιών αυτών και όταν παρατηρούμε ότι υπάρχουν κενά, όταν υπάρχουν προβλήματα, τότε επικοινωνούμε με τα κράτη-μέλη τα οποία δεν υποβάλλουν εγκαίρως τα δεδομένα και αποστέλουμε ουσιαστικά προειδοποιήσει συμμόρφωση ε, στα κράτη αυτά. Μέχρι στιγμή πάντω, ε, σε καμία περίπτωση δεν χρειάστηκε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, εξαιτία απουσία συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολή δεδομένων. Συνήθω όταν υπάρχει κενό συμμόρφωση με την ανταλλαγή επιστολών, το πρόβλημα επιλύεται ανάμεσα στη Eurostat και τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, υπήρχε πάντα μία εθελοντική υποβολή δεδομένων και καταφέρνουμε να πάρουμε στοιχεία από πάρα πολλά κράτη-μέλη. Με την προτινόμενη τώρα, με τον προτινόμενο καονισμό και εφόσον αρχίσει να εφαρμόζεται το 2011, θα έχουμε μία περίοδο μεταβατική δύο ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας πιστεύω ότι θα έχουμε ελάχιστα αιτήματα εξαίρεσης από τον κανονισμό αυτό. Θεωρούμε ότι ήδη από το 2011 και μετά θα αρχίσουμε να συλλέγουμε τα δεδομένα με το σωστό τρόπο από τα κράτη-μέλη, όχι μόνο όσον αφορά την ε, εγκαιρότητα, αλλά όσον αφορά επίσης και την ποιότητα των δεδομένων αυτών. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στις Βρυξέλλες. Καλό ταξίδι πίσω στο Λουξεμβούργο, όπου εργάζεστε, έτσι δεν είναι δεν είναι και πολύ μακριά από εκεί που προέρχομαι εγώ, από τη δική μου την πόλη. Καλή επιτυχία στη δουλειά σας. Voting 9 Στις 9 Οκτωβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή μας και περνάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 6 για την ε, ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σχέδιο ρου, Η κυρία Λιωτάρτα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που διαβάσατε και όλο τον τίτλο. Προσπάθησα να καταρτήσω μια πρόταση για την ενέγισχυση θεμάτων ασφάλειας χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πρινικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια θα αναφέρω μόνο τα αρχικά της πολιτικής αυτής. Το σχέδιο αυτό έχει να κάνει με την ε, προσπάθεια εξέλιψη τέτοιων στοιχείων στην Επιτροπή μας. Πρέπει να εξετάσω τα θέματα που άπτονται της δικής μας ε, αρμοδιότητας. Καλωσορίζω καταρχάς το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει προσοχή στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να αναφέρω ότι θεωρώ ότι η ευθύνη σε ό,τι αφορά τα θέματα τέτοια ασφάλειας καταρχάς είναι στα χέρια των κρατών μελών, αλλά ότι χρειάζεται ασφαλώς συντονισμός και συνεργασία γιατί πολύ συχνά η μόλυνση δεν σταματάει στα εθνικά σύνορα. Και στο παρελθόν λοιπόν έχουμε δει ότι πολλά χάθηκαν επειδή δεν υπήρξε συνεργασία, συντονισμός στα εμβόλια για παράδειγμα για τον ιό της γρήπης πέρσι. Πολλά χρήματα θα είχαμε γλιτώσει αν υπήρχε καλύτερη συνεργασία και θα ήταν πολύ καλύτερα διαθέσιμο και το εμβόλιο από το 1990 και το 2006 ε, έγινε μια ανανέωση της σχετικής νομοθεσίας για τις ε, επιζώτιες. Κρίμα που δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο και για τους ε, ανθρώπινες ασθένειες. Σε ό,τι αφορά τις επιζώτιες θεωρώ να υπάρχει καλύτερο συντονισμό, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ιατρικών υπηρεσιών για παράδειγμα, αλλά και των υποδημών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφιερώνει πολύ προσοχή στην πρόληψη και αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί καταρχάς πρέπει να υπάρχει πρόληψη ασθενειών και επιθέσεων, αλλά κρίμα που δεν αναφέρονται πιο πολλά ως προς την αντίδραση, ως προς τη δράση που θα πρέπει να, να σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να αποτρέψουμε μία επίθεση. Και επίσης πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε μία επίθεση σε ό,τι αφορά ουσίες όπως ο άνθρακας, όπου η περιοχή μόλυνσης είναι πάρα πολύ μεγάλη και ανακαλύπτεται αρκετές ημέρες μετά την επίθεση. Προδίνω λοιπόν στην έκθεσή μου να υπάρξουν σχέδια δράσης και για τέτοιες βιολογικές επιθέσεις. Πάρα πολλές ουσίες μολύνουν το νερό και το έδαφος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσέξουμε την κατάρτιση σχεδίων έγκαιρης, έγκαιρου εντοπισμού των στοιχείων αυτών, αλλά και σε ό,τι αφορά την ε, γρήγορη αποκατάσταση του εδάφους και του ύδατος, γιατί είναι επικίνδυνο να μην ανακαλύπτονται εγκαίρως τέτοιες μολύνσεις και να μην μπορούμε γρήγορα να τις αντιμετωπίσουμε. Επίσης, σε περίπτωση μόλυνσης νερού ή τροφίμων, θα πρέπει να δούμε πώς ε, μπορούμε με καλύτερο τρόπο να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά με το τι επιτρέπεται να φάει και να πιει να τονίσουμε επιτέλους, επί, επίσης, τα μεταφορικά δίκτυα. Χρειάζεται καλή υποδομή για να βοηθούμε ενδεχόμενα θύματα και να αποτρέπεται μόλυνση Θα πρέπει να συμφωνήσουμε επακριβώς τι θα γίνει για τα δίκτυα μεταφορών. Επίσης, με καλύτερο τρόπο θα πρέπει να προσέξουμε τη συνεργασία των ιατρικών υπηρεσιών. Και επίσης, κάτι άλλο που αναφέρω στην χρηματοδότηση είναι η ανάγκη να δίνεται βοήθεια σε ιδιαίτερες ομάδες, σε ηλικιωμένους, σε παιδιά, που χρήζουν ειδική ιατρικής βοήθειας προκειμένου να μην βρίσκονται στο επίκεντρο τέτοιων επιθέσεων. Αν έχουν άλλες ιδέες ενδεχομένω στους συνάδελφοι, ευχαρίστω να τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστούμε την κυρία Λιωτάρ. Chris Davis. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε κάποιες παρατηρήσεις εξ ονόματος του κ. Τζάιες, του συναδέλφου μου, ο οποίος δεν είναι στην αίθουσα. Μου ζήτησε καταρχάς να συγχαρώ την ε, συντάκτρια της γνωμοδότησης, την οποία τη θεωρεί πολύ καλή, πολύ καλά ισορροπημένη, ότι έχει τις απαραίτητες λεπτομέρειες και λαμβάνει υπόψη όλους τους περιβαλλοντικούς και υγειονομικού κινδύνους σε περίπτωση συμβάντων CBRN. Συμφωνεί ότι όντως θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο και να γνωρίζει ότι ο σωστός συντονισμός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανταποκριθούμε ταχαίως στις καταστάσεις. Συμφωνεί επίσης ότι πέρα από την ε, πρόληψη και ε, τον εντοπισμό τέτοιων συμβάντων θα πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και θα πρέπει να έχουμε του απαραίτητου μηχανισμού ανταπόκριση προκειμένου να έχουμε ένα αναρμονισμένο πλαίσιο μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουμε τέτοια συμβάντα το στομότερο δυνατό. Τέλος, ε, συμφωνεί με την αφορά που γίνεται στον μη συντονισμένο υπερβολικό τρόπο που γίνανε οι επενδύσεις για την πανδημία H1N1 και που οδήγησε σε πάρα πολλά δαπάνες στα κράτη-μέλη, δαπάνες οι οποίες δεν ήταν λογικές. Λέει λοιπόν ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε μία έρευνα όσον αφορά τις δαπάνες για την δημιουργία εμβολίων και ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό η Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω κύριος Πρόντι τώρα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σαν σκιώδης εισηγητής θα παρέμβω εγώ από την ομάδα SD. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω τη συνάδελφο εισηγήτρια που κατά την άποψή μου το θέμα το έθεσε με ευρύ και κατανοητό τρόπο. Και κατά την άποψή μου ιδιαίτερα τονίζονται οι βιολογικοί κίνδυνοι όμως και λίγο τα υπόλοιπα. Όπως θα μπορούσαν να αποτελέσουν ε, οι επιθέσεις ε, σε πυρηνικές εγκατεστάσεις ε, αφού θα μπορούσε έτσι να εξαπλαστεί το πυρηνικό υλικό, το ραδιενεργό και αυτό θα είχε ιδιαίτερα σε επιπτώσεις στον πληθυσμό. Θα ήθελα να τονιστεί και το πυρηνικό στοιχείο και το ακτινολογικό, το ακτινοβολίες. Θα τονιστούν και τα δύο. Και επίσης να τονίσουμε την Παρασκευή ε, εμβολίων ε, για τον ιό αυτό, τον HV, και να σας πω ότι αποτέλεσε την πρώτη περίπτωση που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε παρόλο που είχαμε λίγες πληροφορίες και ίσως υποχωρήσαμε, αλλά εντάξει εκ των προτέρων δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε περί τίνος επρόκειται, επρόκειτο και ο κίνδυνος ποιος ήταν. Να τονίσω επίσης ότι δεν αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα καθαρίσουν περιοχές και μια συστηματικού τύπου παρέμβαση ε, για να καθαρίσει σε εισαγωγικά ο τόπος εκεί, η περιοχή εκεί και όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες ε, κινδυνεύουν ε, χημικά και όσον αφορά πυρηνικά και επίσης την πτυχή της ακτινοβολίας. Όλα αυτά απαιτούν μία προετοιμασία που θα πρέπει να γίνεται για κάθε πτυχή του κινδύνου στον οποίο αναφερόμαστε. Αυτά και σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Η κύριε Μαγκουνάιτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω την κυρία Λεωτάρτ, να την ευχαριστήσω για την γνωμοδότησή της, για την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόληψη εξαρτάται από το εκάστοτε κράτος μέλος στον τομέα αυτό. Χρειάζεται ωστόσο και μια κοινή θέση, μια κοινή τοποθέτηση προκειμένου και θεωρώ, συγγνώμη, ότι προ αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Γιατί διανύουμε περίεργους καιρούς και είναι πολύ οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Λόγω αμέλειας των ανθρώπων, αλλά και πολλές φορές. Και λόγω δόλου. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν πρόληψη, όχι μόνο στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλες χώρες και σε άλλα τμήματα του κόσμου, στη Λιθουανία για παράδειγμα, από όπου και προέρχομαι. Το θέμα του CBRN είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, γιατί στην Λουθιανία έχουμε πολλούς τέτοιους κινδύνους, για παράδειγμα τα υπόλοιπα χημικών όπλων σχέδια των γειτονικών χωρών να κατασκευάσουν νέα πυρηνικά εργοστάσια. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει και από σύγχρονες τεχνολογίες. Η αρχή θα πρέπει να είναι η εξής να μην απαγορεύονται συγκεκριμένες τεχνολογίες, αλλά να αυξηθεί το επίπεδο της ασφάλειας. Να συμφωνήσω στο σημείο αυτό με τον κύριο Πρόντι, που μίλησε για την βιολογική μόλυνση, για την διάδοση ενδεχόμενων ασθενειών. Θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και άλλα στοιχεία, θεωρώ. Μου λείπουν από την ανακοίνωση στοιχεία για την αναθεώρηση της τρέχουσας κατάστασης και την εξέταση για την διαπίστωση ενδεχόμενων κενών. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στο σύστημα ασφάλειας, προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες που θα ανακύπτουν. Και να υπάρχει και πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών. ο ορισμός νέων προτύπων ασφάλειας θα οδηγούσε στην αύξηση της ασφάλειας. Δεν θα πρέπει ωστόσο να δημιουργηθούν χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σκοπεύω να υποβάλω κάποιες τροπολογίες και θα πρέπει να συζητήσουμε για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία την οποία και θα υποβάλουμε μετά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θα επιθυμούσε να λάβει τον λόγο. Σας ευχαριστώ Κατερίνα Σβίτσκοβα, ονομάζομαι από την Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι και η συντονίστρια ουσιαστικά για αυτό το σχέδιο δράσης. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης το οποίο διέπει διάφορους τομεί. Θα ήθελα να κάνω κάποιες αρχικές παρατηρήσεις όσον αφορά τα σημεία εκείνα τα οποία έχουν φύγει, Παρουσίες επίσης την οποία παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο τομέας αυτός αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα την αρχή της επικουρικότητας. Γι' αυτό το λόγο το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στην πρόληψη. Και όλα τα σημεία τα οποία θίξετε όσον αφορά την μόλυνση, την απολύμανση, όσον αφορά την ετοιμότητα, όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης, περιλαμβάνονται πραγματικά στο σχέδιο δράσης. Η εφαρμογή όμως αναπόκειται στα κράτη-μέλη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αρχίζουμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε με τα κράτη-μέλη τα συγκεκριμένα βήματα εφαρμογής του σχεδίου δράσης. Και στη φάση αυτή θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα σχόλια τα οποία κάνατε. Και σε αυτή τη φάση θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ότι όντως λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της συμπερίληψης των νέων τεχνολογιών και την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης. Και αυτό το ζήτημα είναι κάτι το οποίο το έχουμε σημειώσει, το έχουμε αναγνωρίσει. Γι' αυτό το λόγο το σχέδιο δράσης ε, περιλαμβάνει και κάποιες προτεραιότητες που βασίζονται στην έρευνα, προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τους κινδύνους, προκειμένου να παρακολουθούμε καλύτερα την εξέλιξη στον τομέα αυτό και προκειμένου να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε και καλύτερα. Η όλη διαδικασία λοιπόν βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι το ότι ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια έκθεση εφαρμογής όσον αφορά το σχέδιο δράσης στα τέλη του 2011. Έκθεση όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογή, σωστή εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης. Επομένως θα έχουμε τη δυνατότητα και στην φάση εκείνη στο 2011 δηλαδή να επανέλθουμε στα σημεία εφαρμογή. Να επιθυμείτε και πάλι το λόγο. Ναι, εν συντομία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που κάναν και την συνάδελφο από τη Λιθουανία. Αν έχει ιδέες για τροπολογίες για τους πυρηνικούς κινδύνους. Θα ήθελα να τις λάβω. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το συζητήσουμε. Για τον κύριο Πρόντι, ο οποίος είπε ότι η έκθεση εστιάζεται κάπως υπερβολικά σε αυτό το κίνδυνο βιολογικής μόλυνσης. Δεν ε, ήταν σκοπός μου αυτός. Ήθελα να αναφερθώ σε όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει πιο πολύ εστίαση στους βιολογικούς κινδύνους, θα ήθελα να το διορθώσουμε αυτό με κάποιες τροπολογίες και ελπίζω να με βοηθήσουν οι συνάδελφοι μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ. Κάτι να υπενθυμίσω. Το μεσημέρι 11 Οκτωβρίου προθεσμία με τη νέα διαδικασία ε, 9 Νοεμβρίου και μετά η ψηφοφορία το Δεκέμβριο του 2010. Έχουμε ακόμα ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Τελευταίο λοιπόν έχει να κάνει με τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρική σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καμερούν για τα δάση το ρόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος ε, Φιλίπ Νίκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την κατάσταση όσον αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αρκετές συναπτυσσόμενες χώρες. Στόχος μου είναι εδώ να σας ενημερώσω, να γίνει μια επικυροποίηση της κατάστασης και να απαντήσω βέβαια και σε ερωτήσεις σας. Ενδεχομένω μπορούν να έχουν να κάνουν περισσότερο με το Καμερούν. Το σχέδιο δράσης το οποίο εγκρίθηκε το 2003 και το οποίο το 2005 μετετρέπει τελικά σε κανονισμό, οδηγεί σε τρεις συμφωνίες. Η μία έχει να κάνει με την Γκάνα, συμφωνία που εγκρίθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο και τώρα έχουμε το Κονγκό και το Καμερούν που βρίσκονται και τα δύο στην τελευταία φάση της διαδικασίας επικύρωσης. Στο διάμεσο διάστημα είχαμε κάποιες άλλες χώρες οι οποίες προσέγγισαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Μαλαισία, Ινδονησία, Κεντρική Αφρική, Λιβερία, Γκαμπόν. Στην Κεντρική Αφρική αυτές οι χώρες λοιπόν. Και σύντομα θα ξεκινήσουν οι πραγματεύσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βιετνάμ ενδεχομένω και με την Γουιάννα και την Παππού Νέα είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις. Με τελευταία ενδεχομένω να ξεκινήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη αρκετέ χώρε οι οποίε ήρθαν σε επαφή μαζί μα και πολλέ διαδικασίε που έχουν ήδη ξεκινήσει. Η βασική ιδέα πίσω από τι εθελοντικέ συμφωνίε εταιρική σχέση είναι απλή. Θέλουμε εδώ πέρα να έχουμε ξυλία η οποία να εξάγεται από ορισμένε χώρε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η ξυλία να συνοδεύεται από μία άδεια, από ένα έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί την νομιμότητα του προϊόντος. Καταλαβαίνετε όμως ότι προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες, δηλαδή πρώτα ένα σύστημα πιστοποίησης ε, των αδειών. Θέλουμε επίσης να πιστοποιεί την νομιμότητα σε όλες τις φάσεις διαδικασίας, όχι μόνο πώς ε, έγινε η συγκομιδή του ξύλου αυτού, πώς έγινε όμως και η παραγωγή του προϊόντος, πώς έγινε η εμπορία του προϊόντος και το καθεξής. Αν λοιπόν τελικό προϊόν φαίνεται να είναι αρκετά απλό, η όλη διαδικασία που οδηγεί στο προϊόν αυτό είναι αρκετά πολύπλοκη. Και θα ήθελα να αφαιρθώ σε τρία επίπεδα πολυπλοκότητας. Πρώτον, η παράνομη δραστηριότητα, δεύτερον, το εμπόριο και τρίτον, η διακυβέρνηση που διέπει τις συμφωνίες αυτές. Όσον αφορά το ζήτημα της παρανομίας, το ζήτημα αυτό είναι περίπλοκο γιατί πολλοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην παρανομία αναφέρθηκα στον τρόπο που γίνεται η συγκομιδή του ξύλου, αλλά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε άλλες περιπτώσεις, στην πώληση του ξύλου, στην εξαγωγή της ξυλίας, θα μπορούσαμε να βρεθούμε στη μεταποίηση του ξύλου. Υπάρχουν πάρα πολλά λοιπόν επίπεδα παράνομης δραστηριότητας που θα πρέπει κάπως να εντοπίζονται από το σύστημα πιστοποίησης της νομιμότητας Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει το στοιχείο αυτό στι θελοντικέ συμφωνίε τερική σχέση. Δεύτερον, το εμπόριο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα πολύπλοκο. Και αυτό γιατί δεν αναφερόμαστε εδώ πέρα σε μια απλή εξαγωγή προς μια, από μια χώρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά με το εμπόριο είναι ότι η ξυλία εξάγεται σε μία χώρα μεταποίησης ή ένα τμήμα της ξυλίας πηγαίνει προς μία κατεύθυνση και το άλλο τμήμα προς μία άλλη. Το να καταφέρουμε λοιπόν να εντοπίσουμε, να παρακολουθήσουμε αυτές τις εμπορικές ροές είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο θέλουμε στις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο να μην παρακάμπτεται. Επίσης σε όλη τη φάση της ε, αλυσίδας εφοδιασμού. Το ξύλο μεταποιείται, παίρνει κάποια άλλη αξία, μεταποιείται σε άλλα προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα στάδια να εντοπίζονται στη, στα πλαίσια της εθελοντικής Συμφωνίας. Τέλος, η διακυβέρνηση, ένα ακόμα πολύπλοκο, ίσως ακόμα πιο πολύπλοκο ζήτημα. Και αυτό γιατί η διακυβέρνηση έχει να κάνει με την εθνική, ακόμα και με την τοπική διάρθρωση που υπάρχει όσον αφορά την χρήση της γης, την ιδιοκτησία της γης, το αν να συμμετέχουν οι αυτόχθονοι πληθυσμοί στη λήψη αποφάσεων ή όχι, ποιο είναι το σύστημα επίσης επιβολής της νομοθεσίας, το οποίο θα μπορούσε να μας εξασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν έχει κάποια πιστοποίηση και ότι όντως πιστοποιείται ως νόμιμο. Όπως βλέπετε λοιπόν η διαπραγμάτευση για τις συμφωνίες αυτές εξελίχθηκε τελικά σε μία συζήτηση και σε μία διαπραγμάτευση για πάρα πολλά και διαφορετικά ζητήματα, τα οποία διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη, μολονότι θα έλεγα ότι η βασική τομή είναι οι ίδιοι. Ουσιαστικά μιλάμε για παράδειγμα για την χρήση και την διοκτησία της γης σε όλες τις χώρες. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να επιληθεί για να αρχίσει να λειτουργεί ένα αποτελεσματικό σύστημα είναι το να καταφέρουμε να κάνουμε μεμονωμένες αποτελεσματικές συμφωνίες με κάθε χώρα. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να εξετάζουμε την περίπτωση κάθε χώρας ξεχωριστά και να έχουμε έπειτα μια πιο προσωποποιημένη προσέγγιση για κάθε χώρα. Κατά αυτόν τον τρόπο η όλη διαδικασία γίνεται λίγο πιο αξιόπιστη και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να συμπεριλάβουμε καλύτερα όλα τα συμβαλώμενα μέρη σε κάθε χώρα, τα οποία μπορεί να μην είναι τα ίδια από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτά είναι, αν τα βασικά, βασικά πλεονεκτήματα, τα βασικά θετικά χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια των εθελοντικών συμφωνιών εταιρική σχέσης ουσιαστικά το ότι έχουμε καταλήξει σε επίπεδο κρατών σε άμεση συζήτηση και διαπραγμάτευση με τα συμβαλόμενα μέρη, με τα ενδιαφερόμενα μέρη που κάθονται στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρομαι εδώ πέρα στον ιδιωτικό τομέα, στην κοινωνία των πολιτών, στις ομάδες αυτόχθονου πληθυσμού και αναφέρομαι θέλετε και σε όλους αυτούς που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα συμφερόντων που έχουν να κάνουν με την ξυλία. Πολύ συχνά έχουμε ακόμα και βουλευτές από τα τοπικά κοινοβούλια στο πλευρό της κυβέρνησης, στην διαπραγματευτική τους ομάδα δηλαδή. Όπως προσπαθούσα λοιπόν να σας εξηγήσω, κάθε εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση είναι διαφορετική και ξεχωριστή, αλλά έχουν όλες την ίδια διάρθρωση, την ίδια δομή και τέτοια στοιχεία. Ξεκινάμε καταρχάς δίνοντας ένα ορισμό για την νομιμότητα. Τι αποτελεί νόμιμο προϊόν με τι θα πρέπει να συμμορφώνεται το προϊόν αυτό προκειμένου να χαρακτηριστεί ως νόμιμο. Βασιζόμαστε βέβαια στα, σε εθνικές νομοθεσίες, στα εθνικά δίκαια και αναφερόμαστε εδώ πέρα στο εργατικό δίκαιο, στο δίκαιο χρήσης και ιδιοκτησίας της γης, σε όλους αστικά αυτούς τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις που μπορούν να πιστοποιήσουν την νομιμότητα που έχει μία εταιρεία για την συλλογή και χρήση της ξυλίας. Ότι δηλαδή η ξυλία αυτή έχει συλλεχθεί με τον νόμιμο τρόπο και ότι μπορούν να την επεξεργαστούν με νόμιμο τρόπο. Στη συνέχεια αναφερόμαστε σε έναν κατάλογο, σε έναν ελάχιστο κατάλογο που αποτελεί τη βάση, αλλά που συνήθως πολλές φορές είναι ανοιχτός και περιλαμβάνει τελικά πάρα πολλά προϊόντα. Έχουμε στη συνέχεια και μια περιγραφή των τεχνικών συστημάτων εξακρίβωσης της νομιμότητας αλλά και της ανοιχνευσιμότητας, Πώς μπορούμε δηλαδή να παρακολουθήσουμε την πορεία του ξύλου από το σημείο στο οποίο κόπηκε ή καλλιεργήθηκε μέχρι το τελικό προϊόν. Επίσης, Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς για την επιτήρηση κάνουν την επιτήρηση αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι όντως λειτουργεί το σύστημα εξακρίβωσης και επιτήρησης. Έπειτα τα μέτρα διαφάνειας στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων ήδη έχουμε μια διαδικασία η οποία θα χαρακτηριζόταν διαφανής. Η συμμετοχή είναι διαφανής, αλλά είναι σημαντικό όλες οι πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις εκχωρήσεις, που έχουν να κάνουν με την ποσότητα ξυλίας που εξάγεται και με το πώς εξάγεται, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι διαφανή, να είναι δημόσια, να κοινοποιούνται, προκειμένου όλα τα συμβαλόμενα μέρη να μπορούν να συμμετέχουν στην εφαρμογή της συμφωνίας. Τέλος υπάρχει και μία κοινή συμφωνία εφαρμογής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αρμόδια κάθε φορά κυβέρνηση, συμφωνία η οποία συνάπτεται προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί με τον κατάλληλο τρόπο η Θελοντική Συμφωνία Εταιρική Σχέση, η VPA. Τώρα το ζήτημα της περιβαλλοντικής ε, βιωσιμότητας συμπεριλαμβάνεται ήδη από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας. Ουσιαστικά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι εθνικές ε, νομοθεσίες ε, ακολουθούν μία βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν συζητάμε την η βιωσιμότητα όπως σας εξήγησα, η αφορία περιλαμβάνεται ήδη στα πολύ αρχικά στάδια της διαπραγμάτευσης της Εθελοντικής Συμφωνίας. Γίνονται κάποιες πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις, υπάρχουν κάποια πολύ ευαίσθητα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κυριαρχία, με τον συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στις διαφορετικές ε, ομάδες. Τα πράγματα δεν είναι απλά και ξεκάθαρα, πάντως η όλη διαδικασία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αποτελεί πάντα μια πρόκληση. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές γίνονται καταρχάς κυρίως μεταξύ των συμμετεχόντων από πλευράς κυβέρνησης, σε εσωτερικό δηλαδή επίπεδο. Διάφορες ομάδες οι οποίε, επαγγελματικέ, για παράδειγμα, οι οποίε δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην κυβέρνηση, καταφέρνουν συμμετέχοντα σε πραγματεύσει αυτές να συμβάλλουν στην οριστικοποίηση της τελικής θέσης της εκάστοτε κυβέρνησης και κατά αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να περάσουν κάποια από τα μελήματά τους στην επίσημη θέση τη χώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, οι σχέσεις αυτές που δημιουργούνται ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, ε, την κυβέρνηση και διάφορους άλλους φορούς και διάφορες άλλες αρχές είναι κάτι το οποίο έπειτα ε, παραμένει και αποτελεί τμήμα τελικά διέπει και τις σχέσεις που δημιουργούνται στην Επιτροπή Εφαρμογής. Και ουσιαστικά η σχέση αυτή η οποία γεννάται στο τραπέζι των πραγματεύσεων διέπει τα έπειτα και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ κυβέρνησης και επιμέρους φορέων στην εκάστοτε χώρα κάθε φορά. Και αν θέλετε αυτό είναι υποφελές και για τις δύο πλευρές. Οι εθελοντικές συμφωνίες τερικέ σχέσεις είναι εμπορικές συμφωνίες. Το εμπόριο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μοχλό προκειμένου να καταφέρουμε να τραβήξουμε το ενδιαφέρον όλων των ενδιαφερομένων, των συμβαλωμένων μερών, με συγχωρείτε, και προκειμένου να καταφέρουμε να πείσουμε τελικά και την κυβέρνηση κάθε χώρας να δημιουργήσει μια εταιρική σχέση με όλους αυτούς τους φορείς σε εθνικό επίπεδο. Ποιες τώρα είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η βασική έχει να κάνει με την διαφάνεια, με το πόσο ξεκάθαρο είναι το νομοθετικό πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η διαφάνεια αυτή. Είναι πολύ σημαντικό η συμφωνία να διέπεται από διαφάνεια, να ξεκάθαρη διάθρωσή τη. Επίσης το ζήτημα της βιωσιμότητας αηφορίας αποτελεί πολλέ φορέ πρόβλημα, γιατί τα συστήματα τα οποία εφαρμόζονται για να συναυθεί η συμφωνία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και μια εθνική νομοθεσία η οποία ενδεχομένως να μην εφαρμόζεται ή θα πρέπει τουλάχιστον να εφαρμόζεται. Επίσης, ξεκινάει ένας διάλογος ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι θεμελιώδης θα έλεγα και είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο οποίο θέλουμε να διατηρήσουμε και στο οποίο προσβλέπουμε. Τώρα το σύστημα πιστοποίησης της νομιμότητας βρίσκεται στην καρδιά των συμφώνιων αυτών και νομίζω ότι θα μπορούσε να συνδυαστεί με την απέτηση για τη διαφάνεια των πληροφοριών και για τη διαφάνεια της διάχυσης των πληροφοριών και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε κατά της διαφθοράς. Πολλές φορές η διαφθορά υφίσταται στις γκρίζες ζώνες της παρανομίας και σιγά σιγά ενδυναμώνεται και γίνεται μία μάστιγα για τις χώρες. Έτσι λοιπόν θέλουμε οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα εξασφαλίζει την διαφάνεια, την πιστοποίηση και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσουμε την ε, διαφθορά. Ουσιαστικά η διαφθορά γίνεται πολύ πιο ορατή κατά αυτόν τον τρόπο στο ευρύ κοινό. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι η επιτυχία των VPA, των συμφωνιών αυτών, αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι όλες οι χώρες με τις οποίες έχουμε περιέλθει στις διαπραγματεύσεις έχουν αποφασίσει όλες να επεκτείνουν την κάλυψη συμφωνίας αυτής πέραν των προϊόντων που εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλυφθούν και όλες οι εξαγωγές τους. Δηλαδή, όλη η ξυλία που φεύγει από το Καμερούν, την, την Κάνα, το Κονγκό, είναι ξυλία η οποία θα διέπεται από ένα σύστημα πιστοποίησης και ανιχνευσιμότητας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, πάντα υπάρχουν τρόποι παράκαμψης της συμφωνίας και γι' αυτό το λόγο Έχουμε πει προς κυβερνήσεις ότι θα πρέπει να βελτιώσουν τις πρακτικές τους όσον αφορά την ε, παραγωγή και την εξογή της ξυλίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσεις για τις εθνοντικές συμφωνίες τερικής σχέσης είναι ιδιαίτερα ευίωνες, πολλά υποσχόμενες. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες χώρες συμμετέχουν σε αυτές και θέλουν να συνάψουν με εμά τέτοιες συμφωνίες. Και θεωρούμε ότι το όλο σύστημα είναι ιδιαίτερα υποσχόμενο. Οι πρώτες άδειες προβλέπονται για το 2011 και πιστεύω ότι αυτό σας βοηθά να καταλάβετε την σημασία της εφαρμογής των συμφωνιών. Δεν είναι μόνο σημαντικό να συνάψουμε τις συμφωνίες, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη, προκειμένου να είναι αξιόπιστες, να είναι αποτελεσματικές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Merci beaucoup, Ευχαριστούμε κύριε Σένη, σας παρακαλώ γρήγορα γρήγορα γιατί θέλουν και άλλοι να λάβουν το λόγο και θα ε, καθυστερήσουμε και έχουν και ένα ωράριο οι διερμηνείς, μην τους ξεχνάμε. I would Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ καταρχάς την, Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε επικριτικοί σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική, αλλά το Flagit πραγματικά αποτελεί ένα υπόδειγμα βέλτιστων πρακτικών για το πώς αντιμετωπίζουμε τους πιο αδύναμους εταιρικούς μας, ε, εταίρους μας. Εφαρμόζουμε τις ευρωπαϊκές μας αρχές με αξιοπρέπεια και με σεβασμό προς τους εταίρους μας. Αναφέρατε ότι οι χώρες αυτές χρησιμοποιούν το εμπόριο, ε, τη, συμφωνία αυτή για το εμπόριό τους στην ξυλία. Υπάρχει το πρόγραμμα Red Plus, το οποίο περιλαμβάνει πληρωμές για συγκεκριμένες υπηρεσίες και από το Red Plus λείπουν κάποιες από τις αρετές του φλεκτ. Κυρίως η συμμετοχική προσέγγιση και η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Είναι σημαντικό και μέσω των διαπραγματεύσεων προσπαθούμε να βοηθήσουμε και το Red Plus να ωφεληθεί από τις εμπειρίες του FLECT και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι πτυχές ε, των υπηρεσιών αυτών. Ευχαριστώ, Κρι Davis, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την παρουσίαση αυτή. Συμφωνούμε, λοιπόν, έχουμε συμφωνίε με τρεις χώρες και καταρχάς οι πρόταση άδειες αναμένεται το 2011. Σας συγχαίρω για το εγχείρημα και πραγματικά σας θαυμάζω πώς καταφέρνετε να αλλάξετε την στάση των χωρών. Δεν μπορώ όμως παρά να είμαι κοινικός η ιδέα με μια συμφωνία να παταχθεί η διαφθορά στο Κονγκό με τους πόρους που έχουμε για την αθηνόμευση, πραγματικά μου φαίνεται επιστημονική φαντασία. Πώς είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει διαφθορά. Για να δούμε τι γίνεται με τις συμφωνίες αλληλείας. Έχουμε υπογράψει συμφωνίες με χώρες οι οποίες απολαμβάνουν ωφέλη, έναντι των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν τελικά. Τα χρήματα αλλάζουν χέρια και τελικά οι ψαράδες παραμένουν εξίσου φτωχοί. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταπιέσουμε, να καταπνίξουμε αυτόν τον κινησμό μας. Υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη η απόδειξη, αν θέλετε, ότι πετυχαίνουμε αυτά που θέλουμε. Και πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτά τα στοιχεία του καταρρεύσει η όλη συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Κανείς άλλος δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Από την Πραβές Επιτροπής μια απαντησούλα, αλλά λίγο λίγο και σύντομα, ε. σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ιδιαίτερα σύντομα. Για το Red Plus. Είναι διαφορετική η λειτουργία του. Πρόκειται για μία πληρωμή, όπως αναφέρεται, για την προστασία του δάσους. Το πρόβλημα με το Red Plus είναι ότι δεν ε, συμπεριλαμβάνει τη διακυβέρνηση ως πρώτο βήμα. Βλέπουμε ότι το FLAG, το FLAGT και το σύστημα διαχείρισης που δημιουργεί αποτελεί, αν θέλετε, το πρωταρχικό στοιχείο για να διασφαλίσουμε ότι οι πληρωμές που γίνονται μέσα στο Red Plus είναι βιώσιμες. Μόνο αν υπάρχει εξ αρχής σωστή διαχείριση και διακυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Γιατί ο κίνδυνος καταστροφής του δάσους συνεπάγεται ότι θα καταργούνταν για παράδειγμα οι πληρωμές μέσα του Red Plus. Άρα θεωρούμε ότι το FLECT αποτελεί τη σωστή βάση για τη διαχείριση του δάσους και για την συνέργεια με τα συστήματα πληρωμών. Το ότι μπορούν να, χρησιμοποιηθούν ε, πληρωμές οικοσυστημάτων, εντάξει, μπορεί. Υπάρχει συμφωνία με την Νορβηγία, για παράδειγμα. Και ως όρος έχει τεθεί να ξεκινήσουν οι Διαπραγματεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει αυτός ο στενός σύνδεσμος, αυτή η στενή σύνδεση, κύριε Ντέιβις, για την διαφθορά. Δεν νομίζω ότι τίφερε θέμα να καταπολεμήσουμε ολοκληρωτικά την ε, διαφθορά. Το θέμα είναι να την εκθέσουμε. Και νομίζουμε ότι έχουμε τις εγγυήσει προκειμένου να αποκαλύψουμε, να φανερώσουμε τη διαφθορά. Είναι η κοινωνία των πολιτών εκείνη που αποτελεί τον πιο ισχυρό μας εταίρο. Θεωρούμε ότι αυξάνοντας την πίεση σε επίπεδο χωρών και στο εξωτερικό, στο εξωτερικό δηλαδή και στο εξωτερικό μιας χώρας, δεν μπορεί κανείς να καταπνίξει την διαφθορά, αλλά μπορεί να περιορίσει τον αντίκτυπό Και εφόσον έχει αποκαλυφθεί η διαφθορά, λειτουργεί το νομικό πλαίσιο και με την κυβέρνηση μπορούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και μαζί με την κοινωνία των πολιτών. Και τέλος υπάρχει και ο ανεξάρτητος έλεγχος. Και να πω στο σημείο αυτό ότι δεν υπάρχει κανένα τέλειο σύστημα αλλά σίγουρα θα δυσκολέψει πιο πολύ τη διαφθορά και σίγουρα θα διευκρινίσει, θα διασαφηνίσει το πώς λειτουργεί το κάθε σύστημα. Είναι πολύ πιο επικοδομητικός τρόπος σε κάθε περίπτωση από το να... Φυσικά υπάρχουν δεσμεύσεις από πλευρά κυβερνήσεων, αλλά πρόκειται για έναν επικοδομητικό τρόπο οικοδόμησης ενός συστήματος το οποίο σέβεται και τα νομικά συστήματα των κυβερνήσεων. Ναι, η πρόεδρος ζητά από τον ομιλητή να συντομεύει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αυτά τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε και Νίκος για όσα μας είπατε. Ήταν πολύ σημαντικά, αρκετά δύσκολο. Αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας, καλή νύχτα σας.